Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Είπαμε ότι σήμερα θα ξεκινήσουμε λίγο αργότερα, 9 και 4. Ευχαριστώ όμως τους συναδέλφους ε, που ήταν εδώ στην ώρα τους. Ε, η συγκήτρια για το πρώτο θέμα ε, είναι εδώ, εδώ και αρκετή ώρα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ηλεκτρονική ψηφοφορία στις 11 και 45. Θα παρακαλούσαμε τους συναδέλφους λοιπόν να φέρουν τις κάρτες για την ψηφοφορία και επίσης να πούμε ότι το θέμα 5 στην ημέρα διάταξη έχει αναβληθεί. Με αυτά λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε από το σημείο 4 που είναι η κατάσταση όσον αφορά το τριμερή διάλογο σχετικά με τον ε, κατάλογο ασφαλών χωρών ε, καταγωγής. Και η συγγήτρια είναι η κυρία Σιλβί Γιόμ. Ο δεύτερο τριμερής διάλογο πραγματοποιήθηκε στι 19 Οκτωβρίου. Σιλβί, σε παρακαλώ αν μπορεί να μα ενημερώσει. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο για να ε, σπάσω και λίγο τον πάγο γιατί κάνει και κρύο σήμερα. Λοιπόν, Έχω συζητήσει τους τριμερείς διαλόγους, τον πρώτο τριμερή διάλογο. Ο, στις 19 Οκτωβρίου έγινε ο δεύτερος τριμερής διάλογος και καταφέραμε να συζητήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα κάποιες προτάσεις και αντιπροτάσεις ε, από τις διάφορες πλευρές και να προχωρήσουμε ε, σε κάποια θέματα, αλλά επίσης και να δούμε και ποια σημεία θα ε, δημιουργήσουν δυσκολίες μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Υπάρχουν τέσσερα βασικά θέματα, θα επαναλάβω για άλλη μια φορά, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Το πρώτο αφορά την εναρμόνιση μεταξύ Ευρωπαϊκού Καταλόγου και Εθνικών Καταλόγων. Ε, να σας υπενθυμίσω ότι εμείς ε, ζητήσαμε να διαγραφούν οι εθνικές ε, λίστες και να έχουμε μόνο έναν Ευρωπαϊκό Κατάλογο των ασφαλών χωρών. Το επιχείρημα είναι, είναι βέβαια από την άλλη πλευρά είναι να υπάρχει συνύπαρξη ε, μεταξύ ε, ευρωπαϊκών και εθνικών καταλόγων. Ε, να σας πω ότι το Κοινοβούλιο έχει σαφή θέση και θεωρούμε ότι είναι ρεαλιστική κιόλα. Εάν διαγράψουμε φυσικά βαθμιδών τους εθνικούς καταλόγους, θα έχουμε και μεγαλύτερη ισχύ της πρότασης. Προτείνουμε μια τριετία. Δεν θα γίνει λοιπόν από τη μια μέρα στην άλλη. Θα υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία και η διαγραφή των εθνικών καταλόγων φυσικά θα έχει πολύ συγκεκριμένες προθεσμίες και ε, όρους για την ε, ε, βαθμιδών κατάργηση των καταλόγων. Ε, το Συμβούλιο θέλει να έχει συνεχή συνύπαρξη μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών καταλόγων, το οποίο θεωρούμε ότι θα αποτελέσει χάος για το μέλλον, διότι δεν θα μας επιτρέψει ε, να έχουμε σύγκληση πρακτικών κυρίως ε, μεταξύ των διαφόρων χωρών όσον αφορά τον, ασφαλών, τον κατάλογο των ασφαλών χωρών καταλογής και φυσικά ελοχεύει και ο κίνδυνος επειδή δεν υπάρχει ε, κάποια αντίθεση σε αυτό, να υπάρχουμε νέους εθνικούς καταλόγους και τελικά θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι εθνικοί κατάλογοι που ο στόχος ε, είναι να τους καταργήσουμε. Ο στόχος λοιπόν του Συμβουλίου σε αυτή την περίπτωση είναι να καθυστερήσει αυτή τη συζήτηση για τη διαγραφή των εθνικών καταλόγων ε, στη συζήτηση για τον κανονισμό για τις διαδικασίες που είναι αυτή τη στιγμή υπό εξέλιξη, αλλά δεν είναι λύση αυτή, δεν μπορούν να ε, καθυστερούν τα πράγματα διότι πρέπει να προχωρήσουμε. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις για να βρεθούν λύσεις για το θέμα αυτό, ε, τουλάχιστον να είμαστε λίγο ικανοποιημένοι, αλλά φτάνουμε, ξεκινούμε από διαμέτρου αντίθετες κατευθύνσεις αν μου επιτρέπετε να το πω. Τώρα, ε, ως προς το επόμενο θέμα, έχουμε προσπάθειες και από τι δύο πλευρέ για να υπάρχουν ουσιαστική πρόοδο. Σε γενικές γραμμές, το Συμβούλιο δέχθηκε να συμπεριλάβουμε και τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, για πηγή ενημέρωσης και να υπάρχει και συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ασύλου για τη διαδικασία. Έχουμε κάποιο πρόβλημα για το ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων ε, στη διαδικασία, για να βρούμε ε, ποια ακριβώς θα είναι η κατάλληλη διαδικασία. Εμείς θέλουμε να υπάρξει πρόοδος βεβαίως, χωρίς όμως να υπάρχει ε, ένας δεν ξέρω πώς να σας το πω, να συμμετέχουν τελικά και να είναι μη κυβερνητικέ οργανώσεις αυτές οι οποίες που θα λαμβάνουν τις αποφάσεις. Εμείς απλώς θέλουμε να συμμετέχουν και να προσφέρουν την εμπειρογνωμοσύνη τους. Ε, προχωρήσαμε, κάναμε κάποιες προτάσεις και περιμένουμε την απάντηση του Συμβουλίου. Το τρίτο σημείο αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εκεί οι συζητήσεις ε, δυστυχώς, ε, λυπάμαι που το λέω, μάλλον θα είναι ιδιαίτερα σύνθετε, διότι οι προτάσεις του Συμβουλίου είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα να είναι λίγο περιφοριακά, καλοπιστικού χαρακτήρα. Ε, στην πραγματικότητα σημαίνει ότι δεν υπάρχει διάθεση για συζήτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα πλαίσια αυτού του θέματος για τους, ε, για τους καταλόγους των ασφαλών χωρών και να το καθυστερήσουν αργότερα για τη συζήτηση για την ε, διαδικασία σύλλου. Εδώ θα είμαι σαφής. Εμείς δεν θέλουμε και σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτή η θέση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Ασφαλών Χωρών δεν θέλουμε αυτή η έννοια των, χωρών, των ασφαλών χωρών καταγωγής να θεωρείται ως κάτι αφηρημένο που δεν έχει σχέση με την πραγματική κατάσταση των ανθρώπων αυτών και των συνεπειών που υπάρχουν για τα άτομα που κάνουν αίτηση ασύλου. Πολλό δε μάλλον, διότι στις προτάσεις που έγιναν από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτές οι νέες προτάσεις που υπάρχουν και συζητούνται, η εφαρμογή της έννοιας ε, της ασφαλούς χώρας καταγωγής και τα διαδικαστικά θέματα θα είναι πλέον υποχρεωτικά. Δεν μπορούμε λοιπόν να ε, θεωρούμε αφηρημένα την έννοια της ασφαλούς χώρας ε, καταγωγής. Είναι λίγο περίπλοκο λοιπόν αυτό το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εμείς όμως ε, ε, τηρούμε επισήμως τη στάση μας και νομίζω ότι οι συζητήσεις πρέπει να συνεχιστούν ακόμα και αν είναι δύσκολες. Και ένα τελευταίο θέμα που συζητούμε είναι ε, ο μηχανισμός αναστολής. Και εκεί υπάρχουν κάποιες προσπάθειες που έχουν γίνει και από τις δύο πλευρές. Να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι το θέμα του μηχανισμού αυτό είναι η δυνατότητα να υπάρχει μια αναστολή για μια χώρα από τον κατάλογο όταν δεν ανταποκρίνεται πλέον η κατάσταση της χώρας στα κριτήρια της ασφαλούς χώρας καταγωγής. Ε, από ό,τι φαίνεται έχουμε τον ίδιο στόχο με το Συμβούλιο, αλλά ακολουθούμε διαφορετικό δρόμο για να επιτύχουμε το στόχο. Ε, ελπίζουμε λοιπόν να υπάρχουν προσπάθειες και από τις δύο πλευρές για να τα καταφέρουμε. Μετά από αυτά τα τέσσερα σημεία στα οποία υπάρχουν ε, διαφωνίες, να πω ότι υπήρχαν ε, κάποια σημεία στα οποία υπήρχε πρόοδος, αλλά από ό,τι ακούσατε υπάρχουν δύο σημεία στα οποία υπάρχει διαφορά και διάσταση απόψεων με το Συμβούλιο. πρέπει να πω ότι στα σημεία αυτά που μας ενδιαφέρουν θα τηρήσουμε αυστηρή στάση και θα προσπαθήσουμε βεβαίως να ε, το συζητήσουμε το θέμα για να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου. Και εδώ επί τη ευκαιρία να ευχαριστήσω και τις τεχνικές ομάδες που μας συνοδεύουν κάθε φορά στις διαπραγματεύσεις και τους κοιόδης συγητές που είναι και παρόντες και πολύ στη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύ πλήρη ενημέρωση. Μία ερώτηση της κυρίας Άντερσεν Μαρτίνα, παρακαλώ. Όχι ακριβώς ερώτηση. Είμαι σκιώδης ε, εισηγήτρια που συνεργάστηκα με την εισηγήτρια και θα ήθελα να γνωρίσω την ε, εξαιρετική δουλειά που έχει να κάνει τους τελευταίους μήνες και θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπε όσον αφορά τις ανησυχίες σχετικά με την ε, στάση του Συμβουλίου, ε, σχετικά με τα βασικά ε, εχέγγυα που θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε κάποια μελλοντική οδηγία ή κανονισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμπεριληφθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και να τηρούνται χωρίς εξαίρεση. Δεν φαίνεται δεν έχουμε καμία εγγύηση ότι θα συμπεριλαμβάνονται σε κάποια μελλοντική οδηγία ή κανονισμό. Και θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό που είπε η συγγήτρια ότι είναι απολύτως απαραίτητο να συμπεριληφθούν στο κείμενο. Δεν θα κάνουμε καμία παραχώρηση στο θέμα αυτό. Και νομίζω ότι και η συγγήτρια και οι άλλοι σκιώδεις ε, θα συμφωνήσουν. Θα επιμείνουν και εκείνοι. Βλέπουμε στην Τουρκία την μαζική σύλληψη 11 βουλευτών. Η Τουρκία με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής χώρα για τους πρόσφυγες, στιγμή που δεν είναι ασφαλής χώρα για τους ίδιους τους πολίτες της. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. να διασφαλίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και να αποτελούν κεντρικό σημείο ε, στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αν δεν έχετε άλλες παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στο σημείο 6. Την ε, έκθεση ε, εκτίμησης κινδύνου της απειλής από το διαδικτυακό οργανωμένο έγκλημα. Έχουμε εδώ μαζί μας ε, τον Στίβεν Βίλσον από το Κέντρο Κυβερναγκλήματος ε, της Europol. Ε, ο κύριος Βίλσον ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά του και βρίσκεται μαζί μας σήμερα για να μας παρουσιάσει την έκθεση. Σας καλωσορίζω λοιπόν. πολύ. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την παρουσίασή σας. Είναι τεράστια η αίθουσα. Γι' αυτό χρειάζεται χρόνος ε, για τα τεχνικά ζητήματα. Ξέρετε, οι ευρωβουλευτέ εδώ επιδεικνύουν μεγάλη ευελιξία. Μπορούν να σα βοηθήσουν και με τεχνικά ζητήματα, αν το επιθυμείτε. Δεν ξέρω αν όλοι βλέπουν την παρουσίαση. Μήπω πρέπει να χαμηλώσουμε τα φώτα λίγο. Όχι, Σιλβί, δεν χρειάζεται να σβήσει τα φώτα δεν ε, εμπίπτει αυτό στα καθήκοντα των αντιπροέδρων. Η κυρία Κιγιόμ, να σας θυμίσω, είναι αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. <laughs> Αλλά προσφέρθηκε να σας βοηθήσει με, την, ε, με τις διαφάνειες. Είμαστε έτοιμοι? Κύριε Βίλσον, σας καλωσορίζω θερμά, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε που προσπαθήκατε να με βοηθήσετε. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα ανέλαβα ως διευθυντής του EC3 και από την προφορά μου θα ακούτε ότι πριν εργαζόμουν στην Σκοτία σε θέματα κυβερνοεγκλήματος. Να περάσω όμως στο EC3. Η πρώτη διαφάνεια εδώ μας δίνει στοιχεία σχετικά με την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος στο κάτω μέρος ε, βλέπετε ότι μιλάμε για εγκλήματα ε, υψηλής ε, τεχνολογίας, πληρωμών και πιο σημαντικό για μένα είναι η προστασία των παιδιών από την σεξουαλική κακοποίηση. Έχουμε την Task Force GCAT που είναι μια ομάδα 12 επιρογνωμόνων από κράτη-μέλη και άλλες χώρες που συνεργάζονται για να ε, καταπολεμήσουν τις πιο ε, σοβαρές ε, περιπτώσεις κυβερνοεγκλήματος όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκοσμίω. 13 υποθέσεις καταφέραμε να κλείσουμε χθε που πριν από 5-6 χρόνια δεν νομίζω ότι θα είχαμε καμία ελπίδα να τις λύσουμε λόγω της πολυπλοκότητάς τους. Επίσης προσφέρουμε στα κράτη-μέλη και βοήθεια εγκληματολογική. Πολλά κράτη-μέλη δεν ε, έχουν το δυναμικό για να αντιμετωπίσουν πολύπλοκες ε, υποθέσεις ε, κυβερνοεγκλήματος και έτσι προσφέρουμε εμείς προστιθέμενη αξία. Πιο σημαντικό τομέα για μένα είναι η πρόληψη του κυβερνοεγκλήματος, διότι είναι πιο σημαντικό να προλάβουμε το έγκλημα από το να πρέπει να κάνουμε τις έρευνες. Επίσης, στρατηγική ανάλυση και οικοδόμηση δυναμικού τα, βοηθάμε τα μικρότερα κράτη-μέλη ώστε να μπορούν να εργάζονται σε πολύ ψηλό επίπεδο όσον αφορά ε, το εγκλήμα. Και τέλος, ε, συνεργασία με ε, τον οικονομικό τομέα και τις κυβερνήσεις στην καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ σήμερα είναι ε, η αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το διαδικτυακό οργανωμένο έγκλημα. Είναι μια έκθεση που ε, εκδίδεται κάθε χρόνο. Και αλλάζει τόσο συχνά το τοπίο ε, στο κυβερνοέγκλημα που πρέπει κάθε χρόνο να δημοσιεύουμε νέα έκθεση, διότι οι περσινές δομές ε, μπορεί να έχουν αντικατασταθεί από καινούριες. Ε, σημαντικό είναι τα στοιχεία που ε, συγκεντρώνουμε από την καταπολέμηση του κυβερνοκλήματος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιούνται στον κύκλο πολιτικής ώστε να δημιουργούνται στρατηγικά σχέδια στα 28 κράτη-μέλη και αυτά να μετατρέπονται σε δράσεις στα, στις επιχειρησιακές δράσεις. Επίσης, εξετάζουμε εάν οι δράσεις μας έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα ε, και αυτό το εξετάζουμε κατά την αξιολόγηση. Οι επιχειρησιακές προτεραιότητες μας ε, για το 2016 ε, συνδέονται άμεσα με την εντολή μας, την εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο και τις άλλες μορφές κυβερνοκλήματος. Αυτό που με έχει εντυπωσιάσει τα τελευταία χρόνια είναι ο τρόπος ε, που οι εγκληματίες ε, λειτουργούν σε πολλά πεδία. Ο καθένας σήμερα έχει στη τσέπη του ένα smartphone ε, και οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται κάθε δυνατότητα που τους δίνουν οι συσκευές αυτές και οι αρχές επιβολής του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπορούν να παρακολουθήσουν τις αλλαγές. Τα βασικά προβλήματα που έχουμε εντοπίσει είναι καταρχάς ε, η κρυπτογράφηση που αποτελεί σημαντική πρόκληση. Πιστεύω ότι η κρυπτογράφηση μπορεί να είναι πάρα πολύ ωφέλιμο εργαλείο για την κοινωνία. Οι περισσότερες ε, εταιρείες που έπεσαν ε, θύματα hacking τα τελευταία χρόνια δεν θα βρίσκονταν στην ίδια περίπτωση αν είχαν χρησιμοποιήσει το εργαλείο αυτό. Ε, θέλουμε λοιπόν να δείξουμε στο κοινό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πόσο σημαντική είναι η κρυπτογράφηση. Η σημαντική πρόκληση για μας όμως είναι η εγκληματική χρήση της κρυπτογράφησης. Πριν δύο με τρία χρόνια έπρεπε κανείς να καταλαβαίνει καλά την κρυπτογράφηση για να τη χρησιμοποιήσει και σωστά. Δυστυχώς όμως ε, έχουν διαδοθεί πολλές ε, καινούριε εφαρμογές ε, που το κάνουν αυτό αυτομάτως. Και έτσι αντιμετωπίζουμε πολύ σημαντικές προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα του εγκλήματος λόγω της χρήσης της κρυπτογράφησης από τους εγκληματίες πιο σημαντική πτυχή για μας, ε, τι αρχές επιβολής του νόμου, είναι να μπορέσουμε να καταστήσουμε καλύτερα τους ε, αξιωματικούς μας, ε, διότι η κρυπτογράφηση τώρα πια είναι τόσο αποτελεσματική που δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με την απλή βία, που χρειαζόμαστε άλλα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Άλλος ε, τομέας ε, όλο και πιο σημαντικός ε, για μας είναι το κυβερνοέγκλημα ως υπηρεσία που παρέχεται. Πριν μερικά χρόνια έπρεπε κανείς να έχει σημαντικό τεχνολογικό εξοπλισμό για τις κυβερνοεπιθέσεις. Σήμερα όμως μπορεί κανείς να αγοράσει την υπηρεσία, δεν χρειάζεται να έχει ο ίδιος τον εξοπλισμό αυτός ε, είναι ένας σημαντικός λόγος που βλέπουμε αύξηση του κυβερνοεγκλήματος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης έχουμε την αυξανόμενη χρήση του σκοτεινού δικτύου Darknet και των κρυφών ε, υπηρεσιών. Και θα πρέπει να καταλάβετε ότι αυτά είναι θέματα που δεν αφορούν μόνο το κυβερνοέγκλημα, αφορούν γενικότερα το έγκλημα. αναφέρθηκα στις σκοτεινές ε, άκορες. Υπάρχουν ε, λοιπόν ε, τρόποι στην, στο διαδίκτυο να κρύψει κανείς, να νομιμοποιήσει στοιχεία κλπ. Και τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται για την διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, δεδομένων και άλλων παράνομων προϊόντων και ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει να προστατεύσουμε τα παιδιά στις περιπτώσεις αυτές και βλέπουμε ότι άλλοι τομείς του εγκλήματος ε, ανοίγονται προς ε, το διαδίκτυο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να εναρμονίσουμε την ε, αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μόνο με ε, γενικότερες έρευνες μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα εντοπίσουμε ε, τον, το μέρος όπου πραγματοποιούνται αυτές οι δραστηριότητες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να ερευνήσουμε τους τομείς αυτούς. Προχωρώ στην ε, εκμετάλλευση παιδιών. Νομίζω ότι αυτή είναι μία από τις ε, μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην, ε, ε, στο τομέα επιβολής του νόμου. Το 2015 και 2016 είδαμε σεξουαλικό εκβιασμό στο διαδίκτυο. Τα παιδιά αναγκάζονται να δώσουν φωτογραφίες δικές τους ή άλλων Ε, ή να, ή να πληρώσουν ε, ή σε μερικές περιπτώσεις και τα δύο. Και δυστυχώς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε δει πολλές αυτοκτονίες παιδιών που βρέθηκαν αντιμέτωπα με τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης, κατάχρηση νομίμων πλατφορμών στο διαδίκτυο. Και αυτό είναι ένας σημαντικός τομέας ε, με τον οποίο ασχολούμαστε. Επίσης, ε, το live streaming της ε, σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Μπορεί κανείς να αγοράσει στο διαδίκτυο την εικόνες κακοποίησης παιδιών. Στις Φιλιππίνες μπορεί κανείς να παραγγείλει σεξ στο διαδίκτυο. και ε, τη μέρα που θα βγω στη σύνταξη θα με ενδιαφέρει να ξέρω τι έχει γίνει σε αυτούς τους τομείς, διότι μπορεί κανείς να κακοποιήσει παιδί από την κρεβατοκάμαρά του στις μέρες μας. Επίσης, ε, στην Europol και στην EC3 ε, σημαντική προτεραιότητα για μας ε, είναι η ταυτοποίηση των ε, θυμάτων. Έχουμε διάφορα εργαλεία στη διάθεσή μας ε, για να μπορέσουμε να αντιστοιχίσουμε φωτογραφίες ε, μεταξύ τους για να συνδέσουμε και έρευνες μεταξύ τους σε διάφορες υποθέσεις. 24, 24 πρόσωπα από τα διάφορα κράτη-μέλη συγκεντρώθηκαν πέρσι για να ταυτοποιήσουν 25 ε, ε, παιδιά που είχαν πέσει θύματα τρομερής ε, κακοποίησης. Και αποκαλύφθηκε ομάδα ε, παιδοφίλων που ε, κακοποίησαν 44 παιδιά τα τελευταία χρόνια. Αυτή για μένα είναι η αξία τη τεχνολογία. Ε, τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή να προστατεύσουμε τα παιδιά μα και μάλιστα όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Και επίση όσον αφορά αυτούς που κακοποιούν παιδιά ε, έχουν ε, εγχειρίδια μεταξύ τους, ε, που μοιράζονται μεταξύ τους σχετικά με το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κρυπτογράφηση και να ξεφύγουν από τις αρχές επιβολής του νόμου. Και μάλιστα εάν ε, κάποιος ε, παραβιάσει αυτές ε, τις οδηγίες ασφαλείας τον απορρίπτουν από το φόρουμ διότι οποιοδήποτε ανακαλυφθεί από τις αρχές αποτελεί απειλή για το σύνολο, το ενός τέτοιου φόρουμ. Επίσης, όσον αφορά το κακό λογισμικό, το malware, είναι κάτι που απειλεί όλους. Ε, παρότι το 2016 είδαμε και πιο στοχευμένες ε, επιθέσεις, ε, έχουν ζητηθεί λίτρα και έχουν χρησιμοποιηθεί κρυπτονομίσματα για αυτό και επίσης αν έχετε μια μικρή επιχείρηση μπορεί να παραβιαστεί το σύνολο της βάσης δεδομένων των πελατών σας. Επίσης είδαμε επιθέσεις ε, στον τομέα της υγείας, ε, τα νοσοκομεία να χάνουν ε, όλα τα δεδομένα τους. Με αποτέλεσμα να μπορεί να πεθάνει άνθρωποι αν δεν ανακτήσουν τα δεδομένα. Είδαμε επίσης επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές. Αυτά λοιπόν αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για μας τους τελευταίους τέσσερις μήνες ε, συνεργαζόμαστε στενά με τον οικονομικό τομέα και ιδιαίτερα με την αστυνομία των κάτω χωρών για να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα όπου όσοι, ε, όσοι έπεσαν θύματα εκβιασμού και τους ζητήθηκαν ελίτρα να μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα του πόσο σημαντικό είναι αυτό για το κοινό. Μέχρι τώρα 25 εκατομμύρια φορές έχουν χακαριστεί ε, ιστοσελίδες. Για να καταλάβετε την κλίμακα του προβλήματος, ε, τα καλά νέα είναι ότι όλα τα κράτη-μέλη συμμετέχουν και πολλοί άλλοι τομείς ε, του οικονομικού χώρου θα συμμετάσχουν. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ε, σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου στην καταπολέμηση του κυβερνοεκκλήματος και περνώ σε ένα πολύ επίκαιρο θέμα, ε, το κυβερνοέγκλημα και τρομοκρατία. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει πολύ σημαντικές επιθέσεις ε, τρομοκρατικές ε, παρόλα αυτά, αυτό αποτελεί απλά θέμα χρόνου. Τα εργαλεία υπάρχουν, η εμπειρογνωμοσύνη υπάρχει σε κάποιες από αυτές τις ομάδες και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου μέχρι να επιτεθούν σε κρίσιμες υποδομές, σε υποδομές ζωτικής σημασίας. Και επίσης σε πρόσφατες ε, επιθέσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είδαμε στοιχεία ε, που συνδέονται με το διαδίκτυο, είδαμε κρυπτογράφηση καθώς και εγχειρίδια ε, για τρομοκράτες ε, σχετικά με το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πιο προηγμένες ε, τεχνικές κρυπτογράφησης για να ξεφύγουν από τις αρχές επιβολής του νόμου. Πάλι υπάρχει ανάγκη για διατομιακή συνεργασία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. το πιο πρόσφατο παράδειγμα του πόσο γρήγορα αλλάζουν τα πράγματα στο κυβερνοέγκλημα. Ε, ήταν ε, οι συγχρονισμένες στοχευμένες επιθέσεις όπου μεγάλος ε, αριθμός υπολογιστών με κακόβουλο λογισμικό επιτίθενται σε έναν ιστότοπο. Με το ίντερνετ των πραγμάτων ε, η απειλή αυτή ε, γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Ε. Πολλά, πολλές συσκευές, άπειρες συσκευές συνδέονται με το ίντερνετ όπως είναι οι εσωτερικές κάμερες ασφαλείας μέχρι το 2020 περιμένουμε ότι 30 δισεκατομμύρια συσκευές θα συνδέονται με το διαδίκτυο και πολλές από αυτές ε, δεν έχουν ε, κανένα ε, μέτρο ασφαλείας. Πριν τέσσερις εβδομάδες στην Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών είχαμε κυβερνοεπιθέσεις και έκλεισαν πολλές από τις μεγάλες επιχειρήσεις και η Λιβερία ε, απεκόπη από το διαδίκτυο λόγω μιας επίθεσης που βασιζόταν σε συσκευές ε, του ίντερνετ των πραγμάτων. Αυτό για μένα γίνεται πολύ σημαντικό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείτε πόσο εξαρτώμαστε ε, στις υπηρεσίες μας, στην καθημερινή μας ζωή από το Internet of Things. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να ε, γίνει επίθεση σε σημαντικές ε, υποδομές. Γι' αυτό σχεδρώνουμε πολλές από τις προσπάθειές μας ε, σε αυτό το θέμα. Είναι μια απειλή η οποία δεν θα εξαφανιστεί και μπορεί κανείς να αποστεθωροποιήσει ολόκληρη χώρα με τις τεχνικές αυτές. Ενιαία στρατηγική μάλλον η στρατηγική για την ε, ε, ενιαία ψηφιακή αγορά προβλέπετε ότι θα, έχει, θα προσφέρει σημαντικό οικονομικό κέρδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τονίζει την ανάγκη για ασφαλή δίκτυα. Εάν ένα δίκτυο δεν είναι ασφαλέ, το κοινό δεν θα τη χρησιμοποιήσει, δεν θα έχει εμπιστοσύνη ε, στο διαδίκτυο και έτσι δεν θα μπορέσουμε ε, να έχουμε το σημαντικό κέρδος που περιμένουμε από το ίντερνετ. Ε, συνεργαζόμαστε στενά με την Ενίζα για να το λύσουμε αυτό και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια των δικτύων εδώ και πολλά χρόνια ε, ε, οι οι αρχές επιβολής του νόμου δεν έχουν ε, συνεργαστεί στενά με την κοινότητα ΣΥΣΕΤ, e αλλά πρέπει να υπάρξει συνεργασία ως συνέπεια του κυβερνοεγκλήματος. Είναι σημαντικό για μας να συνεργαζόμαστε στενά με ε, τις ε, ομάδες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ασχολούνται με προβλήματα υπολογιστών. Και προχωρώ στα συμπεράσματά μας. Οι τομεί σε δράσεις που έχουμε εντοπίσει για το 2016 και 2017 είναι καταρχά η οικοδόμηση υλικού. Αναφέρθηκα ήδη σε αυτό. Στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε τόσο ε, δυνατοί όσο ε, ο πιο αδύναμος κρίκος. Θέλουμε λοιπόν τον κοινό παρονομαστή να τον φέρουμε σε αποδεκτό επίπεδο. Πρόληψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Εάν μπορούμε να, προστατεύσουμε, να προστατευτούμε και να προλάβουμε το έγκλημα, τόσο το καλύτερο. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η νέα γενιά παιδιών καταλαβαίνουν το διαδίκτυο πάρα πολύ καλά. Ε, οι περισσότερες χώρες ε, διδάσκουν γλώσσες ε, στα παιδιά τους. Εγώ νομίζω όμως ότι η κυβερνογλώσσα είναι η γλώσσα του 21ου αιώνα και θα πρέπει να έχουμε ισχυρά εκπαιδευτικά προγράμματα. Πρέπει όμως να έχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα και στις επιχειρήσεις μας και επίσης να εκπαιδεύσουμε και όλους τους αστυνομικούς μας εταιρικές σχέσεις. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να πετύχει από, μόνη, από μόνος το τομέα σε επιβολής ε, του νόμου. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους ε, που μπορούν να μας βοηθήσουν να πετύχουμε ε, τη διαφορά. Τελικά όμως θα πρέπει να κάνουμε έρευνες, θα πρέπει να εξετάσουμε τις συνέπειες του κυβερνοεγκλήματος, θα πρέπει να μπορέσουμε να τη ζήσουμε στα υψηλά επίπεδα εγκληματικότητας για να το πετύχουμε αυτό. Και ε, για μένα ακόμα και περισσότερο από ό,τι σε άλλους ε, τομείς του εγκλήματος ε, το κυβερνοέγκλημα επειδή δεν, δεν σέβεται τα εθνικά σύνορα αποτελεί σημαντική πρόκληση για μας και όσον αφορά την ομοθέσια, θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σκεφτούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά αλλάζουν οι καιροί, αλλάζουν οι τακτικές και θα πρέπει να ε, ασχοληθούμε με την νομοθεσία. Τέλος, έχουμε το πάζλ, το κυβερνοπάζλ. Κοιτάξτε λοιπόν τι έχουμε εδώ. Έχουμε ένα πάζλ εδώ και πολλά χρόνια. Ε, οι, αρχές σε κάθε χώρα αντιπροσωπεύουν αντιπροσώπευαν ένα-δύο κομμάτια. Οι επιχειρήσεις είχαν άλλα δικά τους ε, κομμάτια. Αλλά βλέπουμε ότι οι διάφοροι τομείς αρχίζουν και μοιράζονται μεταξύ τους ε, τις ε, πληροφορίες αυτές και το τμήμα EC3 είναι αποδέκτης των πληροφοριών αυτών και προσπαθούμε να φτιάξουμε το puzzle. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε ποτέ να δούμε την συνολική εικόνα του κυβερνοεγκλήματος. Ε, νομίζω όμως ότι είμαστε σε θέση να διακρίνουμε αρκετούς από αυτούς τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτό, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ε, ας προχωρήσουμε στην ε, τελευταία διαφάνεια. Ήθελα ε, να πω ότι παρότι φαίνεται σαν να έχω μόνο κακά νέα, ε, το διαδίκτυο μας προσφέρει τεράστιες δυνατότητες. Ε, θα ήθελα όμως να σας μεταφέρω το εξής μήνυμα. Είσαστε σημαντικοί άνθρωποι, θα μπορούσαν να πέσουν θύματα και ακόμα και οι οικογένειές σας. Στο Twitter είσαι η 3 Europol κάθε εβδομάδα προσφέρουμε πολύ βασικές πληροφορίες που νομίζω ότι θα κάνουν και εσάς και τις οικογένειές σας πολύ πιο ασφαλείς στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Ορισμένοι συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο για να σας υποβάλουν ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση, λέει ο κύριος Μπόνι μας δώσατε μια πλήρη εικόνα των θεμάτων αυτών. Πρέπει να γνωρίσουμε τη σημασία του έργου της EC3. Έχω ορισμένε ερωτήσεις. Πρώτον, ποια είναι τα νέα μέτρα που λαμβάνει η Europol και η EC3 για να βελτιώσει την πρόληψη προφανώς είναι πολύ σημαντική και επίσης τι θεωρείτε εσείς ότι χρειάζεται, χρειάζεστε για να γίνει η πρόληψη πιο αποτελεσματική. Δεύτερον, αναφερθήκατε στη σημασία της συνεργασίας με άλλους φορείς. Με ποιον τρόπο μπορούμε να τους εμπλέξουμε, να βοηθήσουμε για να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και επίσης για να γίνεται μια αξιολόγηση του κινδύνου σε όλα τα επίπεδα. Από ε, τις επιχειρήσεις, από τις τοπικές αρχές, από τις κυβερνήσεις, πιθανώς ακόμα και από μεμονωμένους πολίτες. Και το ερώτημα μου προς εσάς είναι τι χρειάζεστε για να γίνει ε, πιο αποτελεσματική, για να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των αρχών επιβολής του νόμου. Και τρίτον, αναφερθήκατε στο ζήτημα της κρυπτογράφησης και των προβλημάτων που αυτό δημιουργεί για τις διοπτικές αρχές. Και θα συμφωνήσω, αλλά το ερώτημά μου προς εσάς θα είναι τι, ποιο, ποιο, θα ήταν το πλαίσιο που νομίζετε ότι θα, πρέπει, θα έπρεπε να δημιουργηθεί για να χρησιμοποιείται μεν η κρυπτογράφηση, αλλά με τρόπο αποτελεσματικό που να μην διευκολύνει όμως το έγκλημα. Μετά, για το ζήτημα της ε, ενιαίας αγοράς, Υπάρχει μια προσπάθεια, μια πρωτοβουλία εκεί, αλλά δεν υπάρχει ε, τόσο ε, σωστή συνεργασία, τόσο έντονη συνεργασία όσο θα έπρεπε, έτσι ώστε να υπάρξει μια πλήρης εναρμόνιση όλων των εργαλείων στο πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έπειτα είπατε ότι στο μέλλον μπορεί να υπάρξουν τρομοκρατικές επιθέσει οι οποίες να έχουν χρησιμοποιήσει το κυβερνό έγκλημα πολύ πιο σοβαρά από τη σήμερα. Θα ήθελα να με ενημερώσετε για την αξιολόγηση του κινδύνου που κάνει η Europol. Επίσης, ε, το ζήτημα του ίντερνετ των πραγμάτων. Είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητείται και σε άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Για παράδειγμα, συζητείται στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών, του 5G ή για την, ε, τα τηλεκατευθυνόμενα ρομπότ. Και το ζήτημα που πρέπει να μας αποσχολήσει εμάς εδώ είναι ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε νομοθεσία έτσι ώστε ε, από την αρχή, πριν αρχίσουν να υιοθετούνται και να χρησιμοποιούνται ε, ευρέως αυτές τις συσκευές, να υπάρχει ένα πλαίσιο που να μας εξασφαλίζει. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν ε, λίγους ε, μήνες έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε τι είναι το κυβέρνο έγκλημα και νομίζω ότι κατέστησα σαφές από την παρουσίαση ότι το κυβέρνο έγκλημα δεν είναι κάτι καινούριο, είναι τα παλιά εγκλήματα που με την χρήση ε, ψηφιακών ε, εργαλείων έχουν πολύ πιο ε, εκτενείς ε, συνέπειες. Ε, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται πια να πάω στην τράπεζα να κάνω τη διάρρηξη, να κλέψω τα χρήματα κλπ. Μπορώ να το κάνω από την κρεβατοκάμαρά μου. Πρόκειται λοιπόν για τα ίδια παλιά εγκλήματα, ο, ο τρόπος όμως που διεξάγονται έχει αλλάξει. Η ερώτησή μου είναι, την πρόκληση αυτή μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε αποκλειστικά με τα εργαλεία της ε, αστυνομικής συνεργασίας. Και μπορώ να απαντήσω όχι. Ο συνάδελφος Μπόνι αναφέρθηκε στην ρομποτική. Ε, τι θα γίνει λοιπόν αν κάποιος ε, χακάρει τα ρομπότ αυτά και ξαφνικά ε, ένα ρομπότ κάνει πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να κάνει και μπορεί κανείς να εκβιάσει την επιχείρηση. Επίσης είδαμε παρελειμμένα κλοπή δεδομένων ασθενών και τα νοσοκομεία να εκβιάζονται. Όλα αυτά σίγουρα το βοηθούν και τους ασθενείς. Επίσης, ληστείες σε τράπεζες, το ανέφερα ήδη ερώτηση λοιπόν. Είναι δυνατόν ε, πολλοί να εξακολουθούν να μην είναι προετοιμασμένοι να έχουν ε, ασχοληθεί με την προστασία τους να μην έχουν για παράδειγμα καμία ασφάλεια δεδομένων, να αφήνουν την πόρτα ανοιχτή ώστε οι εγκληματίες ε, εύκολα να μπορέσουν να κλέψουν δεδομένα και όσον αφορά την ε, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών. Παλιότερα, πριν, ε, πάνε, πριν ξεκινήσουν τα παιδιά σχολείο, ε, οι γονείς τους έδειχναν την πρώτη μέρα ποιος είναι ο δρόμος και μετά τα άφηναν να πάνε μόνα τους. Σήμερα τα παιδιά πηγαίνουν με το αυτοκίνητο στο σχολείο και έτσι δεν μαθαίνουν να κυκλοφορούν. Ε, το ίδιο ισχύει με τα ε, ψηφιακά μέσα. Τα παιδιά ε, κάθονται μπροστά στην οθόνη, κανείς δεν τους εξηγεί ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν και αυτό μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά να κάνουν κάτι που δεν θα έπρεπε να κάνουν. Το θέμα της πρόληψης λοιπόν ε, συνδέεται και με ε, τις ε, ψηφιακές ικανότητες. Εσύ τι δυνατότητες ε, βλέπετε για συνεργασία με τα σχολεία, με τους γονείς, ε, με τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών. ώστε ε, τα παιδιά ε, να ε, βλέπουν προσεκτικά, να αντιμετωπίζουν με προσοχή τα, τις προσφορές για επαφή, για παράδειγμα, στο διαδίκτυο. Και επίσης, η κρυπτογράφηση και απλοί πολίτες χρησιμοποιούν ε, την κρυπτογράφηση όχι επειδή είναι εγκληματίες ή έχουν κανένα τεράστιο μυστικό αλλά για να προστατεύσουν την ε, ιδιωτική τους ε, ζωή. Η κρυπτογράφηση όμως χρησιμοποιείται και για εγκλήματα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική πρόκληση. ο οικονομικός τομέας και άλλοι πόσο προετοιμασμένοι είναι όσον αφορά την ψηφιακή προστασία και όσον αφορά την ε, κρυπτογράφηση και ε, πώς μπορούμε να ε, αντιμετωπίσουμε τις οργανωμένες ομάδες εγκλήματος. Ευχαριστώ κυρία Κινίτση. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον ε, καλεσμένο μας ε, για την πλήρη παρουσίαση που μας ε, έκανε για ένα θέμα το οποίο σίγουρα μας ανησυχεί. Μας ανησυχεί όχι μόνο ως Ευρωβουλευτές αλλά ως πολίτες και ως γονείς. Διότι εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε και ίσως ακούστηκε ήδη ότι το έγκλημα είναι το νέο ε, οχυρό του οργανωμένου εγκλήματος, του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος. Ε, το να μπορέσουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μορφή της εγκληματικότητας σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ουσιαστική δέσμευση που θα ε, περιλαμβάνει συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ των διαφορών χωρών. Πολλά σημεία τα έφυξαν οι συνάδελφοι που μίλησαν πριν από μένα, αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ για άλλη μια φορά στο θέμα της πρόληψης. Πολύ σωστά είπατε και η συνάδελφος Σίπελ αναφέρθηκε στο θέμα της πρόληψης, κυρίως για τους ανηλίκους που για άλλη μια φορά είναι η πιο ανυπεράσπιστη σε σχέση με τα εγκλήματα τα οποία διαπράττονται εις βάρος τους ε, μέσω του διαδικτύου. Και ακούστηκε η βία, η σεξουαλική βία, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει και το cyberbullying. Και επίσης ε, ε, και εκεί είχαμε φήματα ε, παιδιά τα οποία αυτοκτόνησαν μετά από αυτή την ε, ε, κακοποίηση, ε, η οποία φυσικά μεγιστοποιείται μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εάν λοιπόν θέλουμε να μάθουμε στους ανηλίκους να χρησιμοποιούν σωστά ε, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και αυτό φυσικά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλό, όπως επεσήμανε και η Μπεργίτη γιατί δεν φτάνουν κατά πάσα πιθανότητα τα σχολεία, ε, πρέπει να υπάρχει και ευαισθητοποίηση των γονέων, οι οποίοι ίσως θα πρέπει να είναι και πιο προσεκτικοί και να γνωρίζουν και αυτοί οι ίδιοι τους κινδύνους του διαδικτύου αυτό ε, το οποίο λοιπόν αναρωτιέμαι είναι τι μπορούμε να κάνουμε από πλευράς πρόληψης όσον αφορά την πάρα πολύ γρήγορη εξέλιξη της τεχνολογίας, την οποία αναφερθήκατε κι εσείς, ε, η οποία μας φέρνει ενώπιον νέων κινδύνων καθημερινά. Είμαστε κατάλληλα εξοπλισμένοι γι' αυτό. Τα πανεπιστήμια, η έρευνα μπορούν να μας βοηθήσουν και θα μπορούσαμε ίσως ε, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ε, διεθνές οργανωμένο έγκλημα σαν αυτό να καταφύγουμε σε εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται σε άλλους τομείς οργανωμένου εγκλήματος και που είχαν καλά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, τους πληροφορίες πληροφοριοδότες, τους whistleblowers. Μπορούμε να έχουμε κάτι αντίστοιχο. Υπάρχει στο Europol ε, ένα κέντρο που να διοικεί αυτά τα πράγματα. Υπάρχει δυνατότητα στη Europol να εργαστούμε και σε θέματα πρόληψης. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως Κοινοβούλιο για να υποστηρίξουμε αυτές τις ε, δεσμεύσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα μέσω του διαδικτύου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκυγιόμ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Στην έκθεσή μας υπάρχουν αρκετές συστάσεις, στην έκθεσή σας, και για την ε, πρόληψη του κυβερνοεγκλήματος, αναφερθήκατε και σε αυτό, και ε, υπάρχουν και προτάσεις για νομοθεσία. Αν δούμε λοιπόν τα διάφορα θέματα που μας απασχολούν όσον αφορά το θέμα των ε, παρισφρήσεων στο Darknet, τα θέματα των επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές, η ποινικοποίηση κάποιων συμπεριφερών. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες επιθυμίες εναρμόνισης κάποιων πρακτικών ε, που αναφέρονται στην εκθεσή σας. Ταυτόχρονα αν είναι σωστές και οι πληροφορίες μου, υπάρχει μία σύμβαση της Βουδαπέστης, όπως αποκαλείται, η οποία μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε σε θέματα ε, κυβερνοεγκλήματος και εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας. Υπάρχει λοιπόν σχέση με αυτή τη σύμβαση, αλλά από ό,τι φαίνεται οι πρακτικές ε, δεν χρησιμοποιούνται πάντα από τα διάφορα κράτη-μέλη. Ε, έχετε κάποιες ε, απόψεις για το πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Ε, ίσως θα μπορούσατε να μας απαντήσετε και αργότερα κύριε Κίνκ, αλλά πραγματικά θα με ενδιαφέρει μια απάντηση από αυτού. Να προσθέσω κι εγώ ρώτησε και η κυρία να αναφέρατε στην παρουσίαση και την ομοθεσία. Υπήρχε και ένα πρόσφατο σεμινάριο για το κυβερνοέγκλημα. Είχαμε εμπειρογνώμονε και μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ασχολούνται με τα θέματα. Και άτομα από τι αρχέ επιβολή του νόμου και αναφέρθηκαν στο πόσο σύνθετα είναι τα πράγματα ή η σύμβαση της Βουδαπέστης αλλά και το, η νομοθεσία στα θέματα αυτά. Σίγουρα μα ενδιαφέρει η κατάλληλη επιβολή αλλά και η ισορροπία ε, μεταξύ ε, επιβολής και κωδικοποίηση για λόγου ε, ε, προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πολλά από αυτά που κάνετε είναι επιχειρησιακή εφαρμογή ε, και φυσικά είναι προστιθέμενη αξία στα όσα κάνουν τα κράτη-μέλη. Τι ε, εννοείται όμως με αυτό, τι θα ήταν πιο χρήσιμο για σας ε, από πλευράς μελλοντική νομοθεσίας και κατευθυντηρίων γραμμών, διότι πολλά από αυτά είναι μάλλον συμβάσεις και δεν είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τι θα ήταν πιο χρήσιμο και τι θα ήταν χρήσιμο, για παράδειγμα, αναφερθήκατε την επίθεση στην Ανατολική Ακτή και στο hacking. Αυτές είναι άμεσες απειλές που μας αφορούν όλους. Τι θα ήταν χρήσιμο λοιπόν από πλευρά νομοθεσίας για να ε, αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, εάν όντω ε, θα έχουμε νομοθεσία και όχι επιχειρησιακή δράση, η οποία ήδη μπορεί βέβαια να ε, υπάρχει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ κύριε και κύριοι. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις με τη σειρά που τη σημείωσα. Καταρχά θα ήθελα να ευχαριστήσω το κυβερνοέγκλημα Λάθος ερώτηση, συγγνώμη, αυτό ήταν από το δεύτερο βουλευτή. Το θέμα της πρόληψης. Πώς βελτιώνουμε αυτά που κάνουμε όσον αφορά την πρόληψη στο λογαριασμό του, του ECC υπάρχουν πολλά περισσότερα. Υπάρχει το EC3 που καλύπτει μια μεγάλη σειρά πληροφοριών για το πώς μπορείτε να προστατευτείτε. Τα καλά νέα σε σχέση με αυτό είναι ότι υπάρχουν κάποια βασικά βήματα τα οποία μπορείτε να λάβετε προκειμένου να προστατευτείτε από απειλές ε, παραδείγματο χάρη, ε, password, να έχετε ενημερωμένο antivirus και να έχετε προστασία από το 80% της απειλής. Αυτό προσπαθούμε να στείλουμε ως μήνυμα στο ευρύ Υπάρχουν πόροι που είναι διαθέσιμοι σε όλα τα κράτη-μέλη, είναι μεταφρασμένα σε παραπλές γλώσσες ε, και προσπαθούμε να στείλουμε ένα κοινό μήνυμα. Τον Οκτώβριο είχαμε το μήνα του ασφαλέστερου διαδικτύου. Ήταν ένας μήνας όπου έγινε μια μεγάλη εκστρατεία ευαισθητοποίηση και δόθηκαν πολλές πληροφορίες διαδικτυακά και υπήρχαν άνθρωποι ε, ε, online που προσπαθούσαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Όλα αυτά είναι μη τεχνικά. Η αλήθεια είναι ότι όταν αρχίζουμε και συζητάμε τεχνικά θέματα, ο κόσμο αρχίζει να μην παρακολουθεί. Και αυτό φυσικά ε, σημαίνει ότι πρέπει να δίνουμε βασικέ πληροφορίε. Το EC3 θέλει να είναι ένα αποθετήριο των πιο ε, επικαιρωμένων πληροφοριών που λαμβάνουμε και από τον κλάδο και από τα πανεπιστήμια και θέλουμε να δούμε τι υπάρχει καλύτερο και να προσπαθήσουμε να τα ε, δώσουμε αυτά. Επίση, προσπαθήσαμε να αναφερθούμε στην ενημέρωση από όλε τι πλευρέ. Όλοι έχουμε ομάδε στη Europol, τα λέμε advisory networks, έχουμε τα πανεπιστήμια, συνεργαζόμαστε με κάποια από τα καλύτερα πανεπιστήμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρησιμοποιούμε τις δομές τους. Ε, ε, μας δίνουν συμβουλές μομοδοτήσεις και σε μεγάλο βαθμό ε, βαθμολογούν κάποια τμήματα για αυτά που βλέπετε στα πανεπιστήμια. Επίσης υπάρχουν δίκτυα του κλάδου, υπάρχουν πάροχοι διαδικτύου, ε, ε τηλεπικοινωνιών, χρηματοπιστωτικό ε, ε, κλάδο και επιχειρήσει διαδικτυακής ασφάλειας. Όλες αυτές είναι ξεχωριστές ομάδες, έρχονται τρεις φορές το χρόνο στη Europol για να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά μας και είναι διαθέσιμοι, μπορούμε να τους καλέσουμε για πληροφορίες πληροφορίες και προσφάτως ε, ζητήσαμε από τους υπευθύνους ασφαλείας για να ε, δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με το malware και ε, ζητήσαμε τη συμβουλή τους. Υπάρχει λοιπόν μια συγχώνευση αρχών επιβολής του νόμου, πανεπιστημίων και κλάδου που είναι πάρα πολύ σημαντική και πιστεύουμε ότι αυτή είναι η λύση. Κρυπτογράφηση. Αναφερθήκατε και στην κρυπτογράφηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ είμαι αναφανδόν υπέρ της κρυπτογράφησης γιατί θα βελτιώσουμε τα πράγματα αν κρυπτογραφούμε όλοι. Αναφερθήκατε όμως και στην κακόβουλη χρήση. Το να προσπαθήσουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε κάτι με τεχνικά μέσα δεν είναι πρακτικό όταν η κρυπτογράφηση είναι τόσο καλή και πιο αποτελεσματική. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να είναι πιο αποτελεσματική. Χρειαζόμαστε λεξικά για να κατανοήσουμε πώς φτιάχνουν τα password του οι άνθρωποι. Ε, να έχουμε περισσότερους πόρους και να εξετάσουμε όχι μόνο τη χρήση των πόρων, αλλά να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση ε, ο διαδικτυακής ε, αποθήκευσης και αποθήκευσης ε, cloud. Και επίσης, όσο προχωράμε στο cloud computing, ε, θα έχουμε λύσεις. Και στην κβαντική, βέβαια, υπολογιστική θα αυξηθεί περισσότερο πύχης και θα έχουμε περισσότερα μέτρα. Δεν έχω κάποια άμεση απάντηση. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να εκπαιδεύσουμε καλύτερα τους υπαλλήλους μας, πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι στον τρόπο με τον οποίο υλοποιούμε κάποια πράγματα και να προσέχουμε. Υπήρχαν αρκετές ερωτήσεις από αρκετά μέλη όσον αφορά την εναρμόνιση της νομοθεσίας και το πώς γίνονται κάποια πράγματα. Για μένα οι αγορές του dark ε, internet είναι η κατάλληλη λύση, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Η ικανότητα λοιπόν να ε, κάνουμε κάποιες ε, επιχειρήσεις με μυστικές. Ε, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα σε κάθε κρατός μέλος και δεν μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα. Αν ξέρουμε ότι υπάρχει ένα ε, στο του Darknet στη χώρα τους, ε, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα κάποιες φορές γιατί δεν έχουν τις δομέ. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει κατάλληλο συντονισμό όπω κάνουμε εμεί στο EC3, να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε το πρόβλημα, να δούμε ποιο είναι ο πλέον αρμόδιο για να το αντιμετωπίσει και από εκεί και πέρα μπορούμε να δούμε τι μπορεί να κάνει το κάθε κράτο μέλο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα πιο αποτελεσματικά. Ε, κάνατε και μία ερώτηση όσον αφορά τι ε, κυβερνοεπιθέσει. Ο συνάδελφος, ο κύριος Ναυρέτια, σας έχει κάνει μία έκθεση για τα θέματα αυτά. Θεωρούμε ότι υπάρχουν δυνατότητες ε, να κλιμακωθούν αυτά τα θέματα. Υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε όλες τις τακτικές που χρησιμοποιούνται για ε, κέρδη, ε, μπορεί να υπάρχουν και για τρομοκρατία. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι όταν βλέπω ότι αυτή τη στιγμή οι ευθύνε ε, του EC3 αυξάνονται, δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στο ε, κυβερνοέγκλημα και στην παιδική εκμετάλλευση. Ε, το 45 με το 50% του προσωπικού μου υποστηρίζει προσωπικό για όλες τις μορφές του εγκλήματος, την τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα και πιθανή προμήθεια και κυκλοφορία πυροβόλων όπλων. Τώρα, για το ίντερνετ των πραγμάτων. Ε, το Κοινοβούλιο ασχολείται με τα θέματα αυτά. Η οικονομική ζωτικότητα του, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται από αυτό. Το ίντερνετ των πραγμάτων λοιπόν αποτελεί τεράστιο πρόβλημα. Εγώ προσπαθώ να το πλωστεύσω. Ασχολούμαι με τον κλάδο και τους ανθρώπους που προμηθεύουν αυτές τις συσκευές. Θα ήθελα να υπάρχουν κίνητρα. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να τιμωρούμε τον κλάδο. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε κίνητρα ώστε να σχεδιάζουν συσκευές οι οποίες θα είναι ασφαλείς από το σχεδιασμό έτσι ώστε να έχουμε ένα κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας για αυτέ τι συσκευέ του ίντερνετ των πραγμάτων, έτσι θα έχουμε προστασία εναντίον μια τεράστια απειλή. Αν δείτε τα στοιχεία που σα έδωσα, 50 δισεκατομμύρια συσκευέ μέχρι τα μέσα του 2020 θα είναι 30 δισεκατομμύρια. Εάν δεν δράσουμε τώρα και δεν αρχίσουμε να σχεδιάσουμε κάποια πράγματα, θα βρεθούμε σε μια ε, κατάσταση μεγάλης αδυναμίας σε 4-5 χρόνια. Τώρα, κάποιες από τις άλλες ερωτήσεις. Αν ε, σχολιάσατε ε, το νέο χειρό όσον αφορά το κυβερνοέγκλημα. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πλέον ε, σύνορα και ορχηρά. Το κυβέρνο έγκλημα ή το έγκλημα το οποίο ε, υποβοηθάται από το κυβέρνο έγκλημα μπορεί να γίνει οπουδήποτε στον κόσμο και να έχει συνέπειε οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Και αυτό είναι τεράστια πρόκληση για μένα. Ρωτήσατε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με το θέμα της πρόληψης. Για μένα αυτό θα έπρεπε να γίνει κάτι το οποίο αφορά και την εκπαίδευση των παιδιών μας από πολύ μικρή ηλικία. Αν δείτε τα παιδιά σα, τα εγγόνια σα, τα νύψια σα, κατά πάσα πιθανότητα θα δείτε τρίχρονα ή τετράχρονα παιδιά να παίζουν με υπολογιστή ή μια έξυπνη συσκευή. Ενστικτοδό αντιλαμβάνονται πώ λειτουργεί. Επομένω πρέπει να υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα του επιτρέψουν να τα χρησιμοποιούν και μάλιστα με ευχάριστο τρόπο. Διδάσκουμε στα παιδιά μα πώ να είναι ασφαλείς στο δρόμο, πώ να κολυμπούν. Ε, ε, νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη απειλή για τα παιδιά μα στο διαδίκτυο. Η ερώτηση λοιπόν και η πρόκληση θα είναι πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην εκπαίδευση των ποδιών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν εξαιρετικοί πόροι, εμείς παρέχουμε αρκετούς και πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, φτάσουμε στα σχολεία στην πολύ νεαρή ηλικία μέχρι και την ε, πλήρη πανεπιστημιακή εκπαίδευση ώστε να έχουμε ταλαντούχους πτυχούχους που θα μπορούν να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους και για την οικονομία. Τώρα, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πολύ γρήγορη αλλαγή τη τεχνολογίας. Εγώ συνεργάζομαι με τον κλάδο και κυρίω ε, συνεργάζομαι με τα πανεπιστήμια. Μέσω της χρηματοδότησης του ορίζοντα 2020 υπάρχουν ε, πρόσβαση σε τεράστια χρηματοδότηση, εξαιρετική χρηματοδότηση, μία από τι καλύτερε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να ε, ε, δούμε και τι γίνεται. Θέλουμε συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, έτσι να επενδύσουμε στα πανεπιστήμια και στον κλάδο και να μπορέσουμε να έχουμε και κάποια θέματα εταιρική κοινωνικής ευθύνης και έτσι να διδάξουμε τους ανθρώπους, να ενισχύσουμε τον κλάδο μας και να βελτιώσουμε και τη δυνατότητα αστυνόμευσης. Ρωτήσατε όσον αφορά τις πιθανούς κινδύνους και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Είναι πολύ ενδιαφέρον ο τομέα αυτός. Ε, συμμετείχα σε ένα πρόγραμμα στη Σκωτία και είδα τα τεράστια ωφέλη που είχε για να αντιμετωπίσουμε το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα στο ύψιστο επίπεδο. Είχαμε κάποιου ανθρώπου που δεν μπορούσαν να του αγγίξει κανεί, δεν μπορούσε να μιλήσει κανεί εναντίον του, αλλά όταν χρησιμοποίησαμε αυτά τα προγράμματα κάτι κάναμε. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την έρευνα του κυβερνού εγκλήματο. Πολλέ φορέ οι εγκληματίε δεν έρχονται από κάποιο ισχυρό εγκληματικό παρελθόν, ε, και αυτό το γεγονός ε, τους δίνει τη δυνατότητα να ε, χρησιμοποιήσουμε ανθρώπους που εργάζονται χρόνια για αυτούς και να ενημερώσουν, να είναι πληροφοριοδότες και whistleblowers. Μπορούν να μας δώσουν πολλές πληροφορίες, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κυρίως για επιθέσεις, για κρίσιμες εθνικές υποδομές, πρέπει, και πολύ σωστά είπατε κι εσείς, να χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες τακτικές που έχουν λειτουργήσει κατά του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας εδώ και χρόνια. Ναι, κάποιες είναι νέε απειλέ, αλλά δεν χρειάζονται μια εκβάθρον νέα ε, ριζοσπαστική προσέγγιση για να τα αντιμετωπίσουμε. Και πάλι ε, υπήρχε και μια ερώτηση όσον αφορά ε, τι γίνεται και κατά πόσον μόνο οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Νομίζω ότι αντιμετωπίσατε αμέσως το, ε, ε, την ερώτησή σας. Πρέπει να υπάρχει σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικό τομέα και συμμετοχή από όλες τις πλευρές. Ακούμε πολλές ιστορίες για τη μη συνεργασία του κλάδου. Εγώ αρχίζω να βλέπω μια ευχάριστη αλλαγή σε σχέση με αυτό. Ο χρηματοπιστωτικό τομέα συνεργάζεται πολύ καλύτερα με εσά. Ο τομέα τη ασφάλεια συνεργάζεται πολύ καλύτερα μαζί μα. Πριν από δύο χρόνια είχαμε μια διάσκεψη στην Europol είχαμε το χρηματοπιστωτικό κλάδο από τη μία και από την άλλη ε, τις αρχές επιβολής του νόμου και ο ένας επέκρινε τον άλλον. Ε, έγινε η ίδια διάσκεψη είχαμε έξι διπλές παρουσιάσεις που έκαναν σε συνεργασία ο χρηματοπιστωτικός κλάδος με τις αρχές επιβολής του νόμου, πώς συνεργάστηκαν, τι αποκόμισαν και τι ωφέλη υπάρχουν. Για μένα λοιπόν αρχίζει να φαίνεται, ε, να διαφαίνεται η δυνατότητα συνεργασίας και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό που χρειαζόμαστε από το Κοινοβούλιο είναι ενθάρρυνση και κίνητρα για τον κλάδο. Δεν χρειάζεται πάντα να υπάρχουν ρυθμίσεις. Τα κίνητρα για μένα τους δίνουν πολύ περισσότερη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικοί. Υπήρχαν και ερωτήσει όσον αφορά την παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση μέσω διαδικτύου. Ε, οι γονεί πρέπει να εκπαιδεύσουν τα παιδιά του, όπω κάνουμε και στον υπόλοιπο κόσμο. Ε, Επίση, οι γονεί θα πρέπει να έχουν και του πόρου για να το κάνουν αυτό. Αυτό που είπα και προηγουμένω. Τα παιδιά πολλέ φορέ μπορεί να είναι πιο. Ε, εύκολα να αντιμετωπίσουν την ε, τεχνολογία. Ε, πιο εξοικειωμένα με την τεχνολογία. Μιλήσαμε με 11χρονα και 12χρονα στη Σκοτία ε, σε ένα πρόγραμμα 12 εβδομάδων και ε, χρησιμοποίησαμε στην πραγματικότητα αυτά τα παιδιά για να πάνε στο σπίτι τους να εκπαιδεύσουν τους γονείς τους και το πιο σημαντικό για μένα τους παππούδες τους ε, οι 70χρονοι που δεν μας καταλαβαίνουν. Αυτό λοιπόν ε, μας επέτρεψε να έχουμε ένα πέρασμα. 11χρονα και 12χρονα παιδιά έδωσαν ε, τον παλμό για τους γονείς τους και για τους παππούδες τους. Τους έμαθαν τα βασικά και τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν από αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια εθνική πρωτοβουλία που έγινε στη Σκωτία και ελπίζω να ε, το αναλάβει και η Ευρωπαϊκή, Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό και να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τα παιδιά για να εκπαιδεύσουν τους μεγαλύτερου. Κύριε Πρόεδρε, και μια τελευταία παρατήρηση για τη δική σας την ερώτηση όσον αφορά την νομοθετική σκοπιά. Ναι, η Σύμβαση της Βουδαπέστης μας δίνει ε, δυνατότητα συνεργασίας ε, και προτείνω να υπάρξει αυτή η συνεργασία. Υπάρχουν ε, ε μεγάλες δυνατότητες και μόνο δύο κράτη-μέλη, ένα ετοιμάζεται να υπογράψει και ένα εκκρεμεί η υπογραφή του. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έχουμε συμμετοχή όλων, αλλά πέραν αυτού εναρμόνιση. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει εναρμόνιση όσον αφορά αυτές τις περίπλοκες, ε, πιθανόν μυστικές έρευνες. Ε, πώς μπορούμε να τα προχωρήσουμε, πώς μπορούμε να ε, ξεπεράσουμε σύνορα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που κάνουμε με τη Eurojust. Υπάρχουν εξαιρετικά ταλαντόχοι νομικοί, οι οποίοι έχουν και τεχνικό υπόβαθρο και μπορούν να μας κατανοήσουν. Και νομίζω ότι η Eurojust έχει πολύ επωφελή ρόλο και μπορεί να βοηθήσει ε, για τις νομικές ε, και πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε εμείς από πλευράς αρχής επιβολής του νόμου και ίσως θα μπορούσαμε με τη συνεργασία αυτή να σας κάνουμε συστάσεις για το τι θα είναι καλύτερο για την νομοθεσία. Νομίζω ότι αυτές είναι οι ερωτήσεις που σημείωσα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Βίλσον για τις λεπτομέρειες απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις των συναδέλφων και για την ε, παρουσίασή σας που γενικότερα νομίζω θα μας δώσει και ιδέες για την συζήτηση που θα κάνουμε αργότερα με τον Επίτροπο. Θα επισκεφτώ την ιστοσελίδα του EC3 για να ε, διαβάσω τα στοιχεία που θα βρούμε εκεί. Είμαι σίγουρος ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ίσως περισσότερο και από εκείνη της Europol. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση σας εδώ, σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Ε, καλή επιτυχία στο, στη συνέχεια του έργου σας. Ευχαριστούμε. Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, ας κάνουμε μια, ένα μικρό διάλειμμα μέχρι τις 10.30, ε, γιατί τότε θα έρθει ο Επίτροπος Κίνγκ. Διάλειμμα στις 10.30 παρακαλώ.

Dear colleagues, we're going to... Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ας συνεχίσουμε τη συνεδρίαση με το σημείο 7. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, μόνο 15 λεπτά. Είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Julian King για τα ζητήματα της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα φροντίσω η εισαγωγή μου να είναι πολύ σύντομη έτσι ώστε να έχουμε χρόνο για την παρουσίαση για τη συζήτηση. Ο επίτροπο Κίνγκα ε, διορίστηκε τον Σεπτέμβριο μετά την ακροασή του και όπως θα έχετε διαπιστώσει ε, ήταν ιδιαίτερα δραστήριος και έχει ήδη κάνει επαφές και συζητήσεις με, με μονομένα μέλη του Κοινοβουλίου της Επιτροπής μας. Θα έχουμε σήμερα λοιπόν τη δυνατότητα να συζητήσουμε στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου για το ζήτημα της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση ο κ. Επιτρόπος και μετά θα γίνει ένας πρώτος γύρος ερωτήσεων. Θα ζητήσω όμως από όλους τους συναδέλφους που θα θέλουν να πάρουν το λόγο για να ρωτήσουν μια ερώτηση να ε, μην ε, τοποθετηθούν, να μην ε, ξεπεράσουν τα δύο λεπτά ομιλίας. Και θα ήθελα ήδη να δω ποιοι συνάδελφοι θα ήθελαν να πάρουν το λόγο για να έχω μια εικόνα. Εάν έχουμε και άλλο χρόνο στη διάθεσή μα θα μπορούσαμε να κάνουμε και δεύτερο γύρο ρωτήσεων Απλώ θα ήθελα να έχω μια αίσθηση από τώρα. Θα μα βοηθήσει και ο επίτροπο στη διαχείριση του χρόνου και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Έχετε το, λόγο. Και καλώ ήρθατε. Ο κ. Κίνγκ, σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Όπως έχω ξαναπεί, θεωρώ τη, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που μου ασκείται πολύ σημαντικό και την παρουσία μου εδώ για να λογοδοτώ εξίσου σημαντική και επίσης θα ήθελα να επαναλάβω ότι οποτεδήποτε ε, θέλετε να μου θέσετε κάποιο θέμα, να με ρωτήσετε κάποιο, ε, για κάποια πληροφορία, μην διστάσετε να έρθετε απευθείας σε επαφή μαζί μου πέρα από τις επίσημες συναντήσεις που θα έχουμε. Ε, το έτος που διανύουμε είναι πολύ σημαντικό ε, μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι. Νομίζω συνεχίζουμε όλοι να θυμόμαστε τις τρομακτικές εικόνες από τους ε, νεκρούς στο εστιατόριο, στον Πατακλάν και βεβαίως τα θύματα και οι οικογένειές τους συνεχίζουν να υφίστανται τις συνέπειες. Υπάρχουν σοβαρά τραυματισμένοι, υπάρχουν άνθρωποι που ε, υπέστησαν ψυχολογικό σοκ. Η ανταπόκριση μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι ήταν εντυπωσιακή ήταν συντονισμένη και αποτελεσματική και θα έπρεπε να αποτελέσει υπόδειγμα για τον τρόπο με τον για αυτό που προσπαθούμε να χτίσουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή μια στρατηγική αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, στην οποία να δίνουμε έμφαση στην ε, βοήθεια προς τα θέματα, η οποία πρέπει να είναι στοχευμένη, να είναι πρακτική να τους δίνει πληροφορίες για τα δικαιώματά τους και ψυχολογική υποστήριξη. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τα θύματα τέτοιων τραγικών ε, τρομοκρατικών επιθέσεων. Ωστόσο, παρά τα βήματα που έγιναν την προηγούμενη χρονιά για να οικοδομήσουμε μια πιο ασφαλή Ευρωπαϊκή Ένωση, η τρομοκρατική απειλή δεν έχει υποχωρήσει, αντιθέτως παραμένει και παραμένει ο κίνδυνος επιθέσεων αδιακρίτων. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε μπροστά μας και προσβλέπω σε, στην ε, διαπραγμάτευση για τρία νομοθετικά κείμενα. Πρώτα απ' όλα τον κώδικα Σέγγεν και την ανταλλαγή στοιχείων ε, για τους ταξιδιώτες, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ε, ιδίω στο πλαίσιο της καταπολέμησης των ξένων μαχητών που επιστρέφουν στις χώρες τους. Επίσης, η οδηγία του Συμβουλίου που θα δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο για την αντιμετώπιση ε, ξένων μαχητών που ε, πηγαίνουν στη Συρία στο Ιράκ. Και το τρίτο είναι η οδηγία για τα πυροβόλα όπλα ε, που θα μας επιτρέψει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι εύκολα προσβάσιμα, δεν θα κυκλοφορούν τα πιο επικίνδυνα πυροβόλα όπλα συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που μετατρέπονται. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε και για να αντιμετωπίσουμε ε, και να βελτιώσουμε μάλλον την πρόληψη και να ε, γίνουμε πιο ισχυρή στον τομέα της καταπολέμησης. Έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο στο επίπεδο της Επιτροπής που είναι το εξή. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ενισχυθεί η ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα. Ήδη ανέφερα τη σημασία που έχουν συστηματική ελέγχη, αλλά επίσης συμπεριληρωματικά προς το προτινόμενο σύστημα ε, ελέγχου στην είσοδο και την έξοδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα θα δημοσιοποιήσει την πρότασή της για ένα πανευρωπαϊκό σύστημα ε, πληροφοριών για τους ταξιδιώτες που επιθυμούν να ε, εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προέρχονται από τρίτες χώρες. Γιατί ένα σύστημα αξιοδότηση. Επίση, θα κάνουμε την, ε, μια αξιολόγηση και θα καταλήξουμε σε προτάσεις για την ε, βελτίωση του συστήματος του πληροφοριακού Schengen, του SIS, το οποίο θα συζητηθεί σε επίπεδο Επίση, Επίσης, ε, αντιμετωπίζουμε γενικότερα προβλήματα, όπως για παράδειγμα η ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων, ζητήματα τα οποία σα απασχολούν και δικαίω. Ε, μια σχετική πρόταση ετοιμάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα δημοσιοποιηθεί τον Δεκέμβριο. Επίση πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα τη χρηματοδότηση τη Τρομοκρατία. Ε, χαίρομαι που σιγά σιγά τίθεται σε εφαρμογή η οδηγία για την καταπολέμηση του ξυπλήματο του μαύρου ε, χρήματο. Από την πλευρά μα, από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε το σχέδιο δράση για την καταπολέμηση τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία και το Δεκέμβριο μια πρόταση για την πολέμηση του ξεπλήματος μαύρου χρήματος, ε, για μια βελτίωση του συστήματος με το οποίο λειτουργούν οι κατασχέσεις και το πάγωμα λογαριασμών. Χρειάζεται λοιπόν βελτίωση της συνεργασίας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά είναι ουσιώδους σημασίας. Το πιο σημαντικό, το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η δικτύωση στο χαμηλότερο επίπεδο, στο οποίο μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει. Ε, για παράδειγμα, αύριο θα οργανώσουμε μια συνάντηση στην οποία θα γίνει μια, ένας απολογισμός και θα συμφωνήσουμε τα επόμενα βήματα. Ε, θα παρευρίσκονται και εκπρόσωποι του κέντρου Αριστείας ΡΑΝ, το οποίο θα μας παρουσιάσει το έργο του και θα δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα δικτύο, ένα αποθετήριο, ένα σύστημα με το οποίο τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα, οι ειδικοί των κρατών μελών θα έχουν τη δυνατότητα να αντελάσσουν με τους συναδέλφους τους βέλτιστες πρακτικές και να εξ... Ε, βρούμε τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση των νέων, που είναι και το αντικείμενο του αυριανού συνεδρίου. Όπως εσύ είπα πρέπει να ενισχύσουμε τις ικανότητες άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συμπεριλαμβάνει την ενίσχυση υπηρεσιών της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τις τελευταίες εβδομάδες ε, επισκέφθηκα ε, υπηρεσίες όπως την Europol, την Eurojust, την EULISA, υπηρεσίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και φορείς με τις οποίες συνεργαζόμαστε και έχω εντυπωσιαστεί από τη συνεισφορά τους και από την ποιότητα του έργου τους θα προσπαθήσω να τους υποστηρίσω ζω όσο περισσότερο μπορώ διαρκώς η Europol έχει στη διάθεση της πια λειτουργεί πλέον σε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο της δίνει τη δυνατότητα να είναι πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της τροποκρατίας, με το κέντρο ε, το καταπολέμηση της τροποκρατίας που δημιουργείται. Θα πρέπει επίσης να δούμε πώς θα ενισχυθεί ο ρόλος της Eurojust στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Έχει γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τους ε, υπουργούς στο Συμβούλιο Υπουργών του Λουξεμβούργου τον προηγούμενο μήνα και βεβαίω θα ήθελα να ξέρω, να γνωρίσω και τις ε, απόψεις του Ευρωκοινοβουλίου. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του χαρτοφυλακίου μου είναι η εφαρμογή των, αποφάσεων. Δεν μιλώ για τις διαδικασίες επί παραβάση τις οποίες θα μπορούσε να ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι ο στόχος μας να συλλέξουμε πρόστιμα, αν και βεβαίως δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το αυτή τη διαδικασία όταν είναι απαραίτητο. Το ζήτημα είναι να είναι ε, διατεθειμένα τα κράτη-μέλη να, να εφαρμόζουν τις αποφάσεις που από κοινού λαμβάνουμε. Και προετοιμάζουμε ένα σχέδιο δράσης ε, το οποίο θα καλύπτει την περίοδο μέχρι την άνοιξη του 19 για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων στο τομέα της δημοκρατίας. Τώρα, σε σχέση με την ομάδα υψηλού επίπεδου εμπειρογνωμόνων για τα πληροφοριακά συστήματα και τη διαλειτουργικότητα, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η ποιότητα των δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους οι συνοριοφύλακες και οι αρχέ. αρχές. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ε, μια διαπαφή, ένα interface ε, για τι αναζητήσει, το οποίο να είναι μοναδικό και ενιαίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς αυτό βεβαίως να αλλάζει τους κανόνες που διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση των δεδομένων. Αλλά να υπάρχει ένα σύστημα με το οποίο όλες οι διοκτικές αρχές να μπορούν να ε, ε, ε, αναζητούν αυτά τα στοιχεία. Ήδη τον Δεκέμβριο θα γίνει η πρώτη συζήτηση για αυτό το θέμα, με τη συνεισφορά των εμπειρογνωμόνων από όλα τα κράτη-μέλη, που σημαίνει ότι αργότερα θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε και μαζί. Όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, στην πρώτη μας συνάντηση είχα δεσμευτεί ότι θα γίνει μια συνολική αξιολόγηση των αποτελετικών που έχουμε για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2011 είχε εγκρίνει ένα ψήφισμα το με το οποίο ζητεί μια τέτοια αξιολόγηση και είχε θέσει και πολύ φιλόδοξους στόχους. Εγώ από την πλευρά μου ήθελα να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα και για την έλλειψη αποτελεσματικότητας των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και να έχουμε ένα έγγραφο στη διάθεσή μας για να το συζητήσουμε την αρχή της, στην αρχή του επόμενου έτους. Σε αυτή την αξιολόγηση βεβαίως θα συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με άλλους θεσμικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, θα οργανώσουμε συναντήσεις και εργαστήρια. Όλα αυτά θα γίνουν τους επόμενους μήνες. Αυτά από την πλευρά μου. Σας ευχαριστώ για την πρώτη συσοχή σας και όπως είπα και πάλι είμαι ιδιαίτερος ευτυχής που έχουμε την δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πολύ μακρύ κατάλογο ομιλητών. Θα κλείσω τον κατάλογο και θα σας παρακαλέσω να περιοριστείτε στα δύο λεπτά για να ακούσουμε τις απαντήσεις ε, το, του Επιτρόπου. Θα ξεκινήσουμε από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, που ήρθατε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ και για τις προσπάθειές σας τους τελευταίους μήνες ε, για να βελτιώσετε την κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα ακούμε ανθρώπους που εκμεταλλεύονται τους φόβους ανθρώπους και προσπαθούν να συνδέσουν την μετανάστευση με την τρομοκρατία. Είναι δύο ξεχωριστά θέματα τα οποία απαιτούν και ξεχωριστή προσέγγιση και ξέρω ότι και εσείς εσημερίζεστε τη θέση αυτή όπως και πολλοί συνάδελφοι στην Επιτροπή μας. Παρότι αυτό είναι ένα φύγμα στο οποίο θα πρέπει να αντισταθούμε, θα κρύβαμε το κεφάλι μας ε, στην άμμο και θα επιτρέπαμε ε, στα λαϊκιστικά κινήματα να αναπτυχθούν ε, εάν αγνοούσαμε την πραγματικότητα ότι η μετανάστευση έχει κάποιους κινδύνους στους οποίους θα πρέπει να απαντήσουμε ως νομοθέτες. Υπάρχουν φόβοι όσον αφορά την κατάσταση της ασφάλειας και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν τα απαραίτητα στα εξωτερικά σύνορα για να διασκεδάσουμε αυτούς τους φόβους. Ε, και είναι κρίσιμη σημασία ε, το σύστημα ε, αίτιας για τις πληροφορίες και την αδειοδότηση των ταξιδιωτών. Αυτό λοιπόν θα είναι ένα σύγχρονο και απαραίτητο εργαλείο. Ταυτόχρονα, όσο πλησιάζει η επέτειος των επιθέσεων στο Παρίσι, θα πρέπει να φροντίσουμε οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου μας και αυτοί που μπορούν να ε, μοιράζονται δεδομένα, ε, να σέβονται την προστασία των δεδομένων και να φροντίσουμε να είναι συμβατά μεταξύ τους ε, τα συστήματα. Απέχουμε πολύ από αυτό και θα πρέπει οι πολίτες μας να έχουν εμπιστοσύνη στα συστήματα που εφαρμόζουμε στα εξωτερικά μας σύνορα για να είμαστε ένα βήμα μπροστά από τα τρομοκρατικά δίκτυα. Νομίζω ότι οι προσπάθειε τη Επιτροπή αποτελούν πολύ καλό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μετά από τις τρομοκρατικέ επιθέσεις πάντα αλλάζει η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια και υπάρχει ανάγκη πότε πότε να ελέγχει κανείς. Υπάρχουν μέτρα που εφαρμόζονται τα οποία δεν είναι πια απαραίτητα. Είναι απαραίτητο να έχουμε ενισχυμένη και πιο αποτελεσματική χρήση των εργαλείων που ήδη έχουμε και μόνο τότε μπορούμε να αποφασίσουμε αν είναι απαραίτητο ε, να θεσπίσουμε νέα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε νέε προκλήσει. Εμείς εδώ ξεκινήσαμε από το τρίτο βήμα. Μιλάμε για νέα μέτρα, όπως είναι το PNR. Μετά λοιπόν από τις πρώτες επιθέσεις πέρσι διαπιστώσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών ε, και εντός των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών πιο σημαντικό. Ε, μάθαμε από αυτά, δεν είμαι βέβαιη. Η ανταλλαγή πληροφοριών ε, εντός δεδομένων και μεταξύ των κρατών μελών δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει σημαντικά. Ε, μπορούμε λοιπόν να ελέγξουμε όσον αφορά την αστυνομία στα κράτη-μέλη ε, έχουν το απαραίτητο δυναμικό και τις απαραίτητες δεξιότητε για να αντιμετωπίσουμε τις απειλές. Όσον αφορά την ανταλλαγή των πληροφοριών, χρειαζόμαστε μια περισσότερη εις κατανόηση των διαφόρων δομών και των τρόπων που ε, εργάζεται η αστυνομία στα διάφορα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σύστημα σαν το Εράσμους μεταξύ αστυνομικών, όχι μόνο σε υψηλό επίπεδο, αλλά και των ε, αστυνομικών που κάνουν την ε, κανονική καθημερινή δουλειά. Και χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία και περισσότερε κοινέ ομάδε ερευνών για να έχουμε καλύτερη κατανόηση και καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά την καθημερινή πρακτική εργασία. Είπατε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών. Το θέμα είναι πόσο έχουμε προχωρήσει στο θέμα αυτό και μπορούμε πράγματι να αποδείξουμε ότι νέα μέτρα όπως είναι το PNR Εσείς είπατε ότι θα φροντίσετε για την εφαρμογή, αλλά η δική μου ερώτηση είναι Είμαστε ακόμα βέβαιοι ότι θα επιφέρει προστιθέμενη αξία αυτό το σύστημα αυτό. Ε, δεν είμαι βέβαιη και κλείνω λέγοντας ότι τα κράτη-μέλη φαίνεται να μην το πιστεύουν διότι δεν ε, φαίνεται να βιάζονται να ε, εφαρμόσουν το μέτρο αυτό το οποίο ζήτησαν τόσο επιτακτικά. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ε, βελτιώσουμε πρώτα τα παλαιότερα μέτρα που έχουμε προτού πανίσουμε ένα σωρό χρήματα πάνω σε αυτό το μέτρο. Από το ECR παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κατά τον προηγούμενο διάλογό μας ε, σας ε, ζήτησα τις απόψεις σας ε, σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία για τα πυροβόλα όπλα. Τώρα που, που πραγματοποιείται ο τριμερής διάλογος θα ήθελα να σας ξαναρωτήσω και θα ήθελα πιο συγκεκριμένη απάντηση από το ότι απλά θέλετε ένα δίκαιο και ισορροπημένο αποτέλεσμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να επιμένει σε πλήρη κατάσχεση και απαγόρευση για τα ημιαυτόματα ε, όπλα για αθλητικές δραστηριότητες, παρότι αυτό έχει επικριθεί σημαντικά και ε, στο ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και παρότι καμία εγκληματολογική έρευνα δεν φαίνεται να δείχνει ότι αυτό το είδος όπλων το οποίο αποκτάται νόμιμα αποτελεί απειλή για την ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αρχίσει να σέβεται τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καλή νομοθεσία από τις αρχικές ε, σύντομες παρατηρήσεις σας. Ε, μου δόθηκε η εντύπωση ότι μάλλον νιώθετε ενθουσιασμό για την ε, πρόταση αυτή της Επιτροπής. Ελπίζω όμως να είναι ψευδής η εντύπωση μου αυτή. Ευχαριστώ. Και η κυρία Βίξτρομ από την Άλτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ μαζί μας σήμερα. Ε, χαίρομαι πολύ που ήδη έχετε ξεκινήσει τον διαφρομένο διάλογο με την Επιτροπή μας. Είναι κάτι πολύ απαραίτητο και είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, για μας το χαρτοφυλάκιο. Μπορεί να ακούγομαι σαν ε, χαλασμένος δίσκος, αλλά θα ήθελα να ξαναθέσω το ίδιο θέμα. Ανταλλαγή πληροφοριών ως απαραίτητο στοιχείο για μια αποτελεσματική ένωση ασφαλείας. Χαίρομαι που ε, συνάδελφοι όπως ο Ρομπέρτο Μέτσολα ήδη το ανέφεραν. Είναι σημαντικό, η Ρομπέρτα Μέτσολα, είναι ε, σημαντικό να, ε, να γίνεται σωστά η ανταλλαγή πληροφοριών. Και δεν μιλάμε για την ε, κοινή βάση δεδομένων, αναφερόμαστε απλά στην ε, ανταλλαγή ε, συγκεκριμένων ε, πληροφοριών από το ένα, κράτος, ένα μέρος στο άλλο και τη συγκέντρωση των πληροφοριών αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, στο τέλος της παρέμβασής σας αναφερθήκατε στην εφαρμογή της οδηγίας PNR και λυπούμεθα για την ε, ε, κάπως ε, αδύναμη ανταπόκριση των κρατών μελών. Ε, χαιρόμαστε που αποτελεί προτεραιότητα για εσά αυτή η οδηγία. Όλοι όμως γνωρίζουμε ότι η προστιθέμενη αξία της δημιουργίας 28 διαφορετικών βάσεων δεδομένων ε, θα είναι περιορισμένη, αν όχι ε, ανύπαρκτη. θα πρέπει προορατικά να γίνεται ανταλλαγή δεδομένων PNR ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αυτή ήταν μια από τις προτεραιότητες μας ε, κατά τις διαπραγματεύσεις. Ε, πρέπει όμως ε, να διαπιστώσουμε υποκρισία από πλευράς του Συμβουλίου. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, τι συγκεκριμένες δράσεις σκοπεύετε να αναλάβετε κατά την εφαρμογή της οδηγίας PNR για να διασφαλίσετε οι απαραίτητε πληροφορίε να ανταλλάσσονται με τον ε, βέλτιστο και αποτελεσματικό τρόπο ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ε, επίσης, η ομάδα μου έχει προτείνει περαιτέρω μέτρα πάνω στο θέμα αυτό ε, που έχουν να κάνουν με την υποχρέωση ερευνών και όσον αφορά τη μελλοντική οδηγία για την ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ελπίζω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να έχουν ε, ε, θετική στάση απέναντι σε αυτές τις προτάσεις και τις δηλώσεις τους να τις μετατρέψουν σε πραγματική πράξη. Κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι θα είναι απαραίτητη η βοήθειά σας. Ευχόμαστε λοιπόν το καλύτερο τις ε, συνομιλίες με τα κρατη πάνω στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Κορνίλια Έρνστ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κίν, καλώς ήρθατε. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο θέματα. Από ριζοσπαστικοποίηση. Θυμάμαι την δήλωσή σας ότι είναι σημαντικό να αναλυφθούν μέτρα για το θέμα αυτό και η ερώτησή μου είναι εσείς ε, τι προτείνετε. Ποιες ε, είναι οι, ε, στρατηγικ... στρατηγικές σας προτεραιότητες. Πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα ε, και κατόπιν να προτείνουμε μέτρα, αλλά δεν μπορέσαμε να λύσουμε το θέμα. Και επίσης εξέταση των μέτρων ασφαλείας. Είναι πολύ θετικό το ότι θέλετε να το κάνετε αυτό το πρώτο εξάμεινο το 2017, να εξετάσετε, να αξιολογήσετε τα μέτρα ασφαλείας. Θα ήθελα όμως να ξέρω από εσά ε, πώς θέλετε να το κάνετε αυτό, με βάση ποια κριτήρια. Και είσαστε διατεθειμένος επίσης να θεσπίσετε μέτρα ασφαλείας ε, ε, παράνομα, για παράδειγμα, έχουμε την ε, συμφωνία PNR με τον Καναδά, που επικρίθηκε από το δικαστήριο. Είσαστε διατεθειμένος ε, να δεχτείτε τις συνέπειες να εξετάσετε με κριτικό μάτι την ε, συμφωνία PNR της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τις αποσύρετε σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ότι δεν είναι σύνομες. Και επίσης, τα μέτρα αυτά ε, ενεργούν αθρηστικά, αλλά είσαστε διατεθειμένος να τα αποσύρετε σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι δεν είναι αποτελεσματικά ή σε περίπτωση που απορριφθούν από το δικαστήριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι διαφωνούμε όσον αφορά το πώς θα πετύχουμε την ασφάλεια της Ευρώπης ε, και εσείς μας δώσατε πολλά παραδείγματα σχετικά με το πώς μπορούμε να ελέγξουμε τα εσωτερικά και εξωτερικά μας σύνορα. Εάν όμως εξετάσουμε τον ε, μακρύ κατάλογο τρομοκρατικών επιθέσεων ε, στην Ευρώπη, βλέπουμε ότι οι περισσότεροι τρομοκράτες είχαν ευρωπαϊκά διαβατήρια. Έχουμε εσωτερικό πρόβλημα που έχει να κάνει με τις κοινωνίες μας. Μιλάτε για ανθεκτικότητα της κοινωνίας, αλλά η ανθεκτικότητά μας θα πρέπει να έχει να κάνει με την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και να δώσουμε μια προοπτική στους ανθρώπους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλουμε ασφάλεια μόνο κατά τη διέλευση των συνόρων, δεν νομίζω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα, ούτε ότι θα γίνουν πιο ανθεκτικέ οι κοινωνίε μα. Ε, θα ήθελα λοιπόν να μου αναπτύξετε την πρότασή σα ε, για την καταπολέμηση τη ριζοσπαστικοποίηση. Δεν άκουσα να λέτε τίποτα για την κρυπτογράφηση, ενώ κατά την ε, ακρόασή σα συζητήσαμε το θέμα αυτό. Αυτό τι σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκαταλείψει την ιδέα ε, σχετικά με τα κρυπτογραφημένα τεκμήρια. Σας παρακαλώ να μας τα εξηγήσετε αυτό. Και ενώ επικροτούμε αξιολόγηση των πολιτικών κατά της θερμοκρατίας, θα θέλαμε να συμμετέχουμε και σε αυτές ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη διαμόρφωσή τους. Και να προχωρήσω τώρα στην οδηγία κατά της νομοποίησης παράνομων εσόδων. Ως ε, συνεισηγήτρια της στην ε, ΛΥΠΕ, ε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η έκθεση αυτή ε, μεταφράζεται, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε με την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στην πέμπτη οδηγία για την νομοποίηση παρανομών εσόδων διότι ε, φαίνεται να μην έχουμε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το τι θα είναι αποτελεσματικό και έχουμε ζητήσει από διάφορους να μας δείξουν, αλλά δυσκολευόμαστε στο θέμα αυτό, διότι ε, δεν έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα τα δεδομένα ε, στα οποία δεν δίνεται πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προτού να έχω περισσότερες ε, πληροφορίες, δεν νομίζω ότι το να παρακολουθούμε τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αποτελεί και λύση για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε, αν θέλετε να απαντήσετε πρώτα στον πρώτο γύρο ερωτήσεων και μετά θα ακούσουμε το δεύτερο γύρο, αφού απαντήσετε στους συντονιστές. Ναι, να προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις ε, ε, ευρύ το φάσμα τους. για το θέμα της μετανάστευσης και της τρομοκρατίας. Νομίζω ότι όλοι, ελπίζω μάλλον όλοι να συμφωνούμε για το πώς ε, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τα θέματα αυτά. Υπάρχουν θέματα όπως η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, θέματα τα οποία διαφέρουν και είναι ξεχωριστά από τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την τρομοκρατία. Και αν ε, συμπτύξουμε τα δύο, τότε ουσιαστικά κάνουμε το προπαγανδιστικό έργο του, ε, και ε, δίνουμε και ε, τροφή ε, σε λαϊκιστικά κινήματα τα οποία θέλουν να εκμεταλλευτούν την πραγματική τρομοκρατική απειλή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να τα συνδυάσουν με τις μεταναστευτικές ροές. Υποστηρίζω λοιπόν ακράδαντα αυτό το οποίο έλεγε η κυρία Μέτσολα επ' αυτού και πιστεύω ότι πρέπει συνεπώς στα μηνύματα που αποστέλουμε να κάνουμε αυτή τη διάκριση. Πέραν αυτού γνωρίζουμε ότι κάποιοι ε, οι οποίοι έχουν ε, ε, συνεργαστεί με τον ISIS και προσπαθούν να μας ζημιώσουν, να μας κάνουν κακό, έχουν επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιούν τις ίδιες διαδρομές που χρησιμοποιούν και οι μετανάστες. Επομένως θεωρώ ότι έχει σημασία το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει μια σαφής περιγραφή των μέτρων που λαμβάνονται προκειμένου να ενισχύσουμε τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων μας ε, στα σημεία εισόδου. Διότι αυτό είναι τμήμα της απάντησης ε, προς αυτούς που προσπαθούν ε, ψευδώς να συνδυάσουν θέματα μετανάστευσης και τρομοκρατίας. Αν ότι υπάρχουν αποτελεσματικοί έλεγχοι στα σημεία εισόδου μέσω της χρήσης ε, πλέον της ε, ε, ακτοφυλακής και συνοριοφυλακής, κυρίως στην Ελλάδα και στην Ιταλία, αρμοδιότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, των αρχών τους και φυσικά επικροτούμε τις προσπάθειες που κάνουν. Η Ιταλία έχει αυξήσει σημαντικά το ρυθμό με τον οποίο καταγράφει και λαμβάνει δακτυλικά αποτυπώματα των ε, ανθρώπων που φτάνουν στα σύνορα. Και αυτά φυσικά συνδυάζονται και με τα όσα κάνει η Europol επιτόπου και στην Ελλάδα και σύντομα και στην Ιταλία για να βοηθήσει και να υποστηρίξει τις εθνικές αρχές όπου απαιτείται και όπου αιτιολογείται να κάνουν και σε δεύτερο βαθμό ελέγχους εάν κάποιος από τους αφιχθέντες ε, δίνει λαβή για παρακολούθηση ή για κάποιον επιπλέον έλεγχο. Πέραν αυτού υπάρχουν και μέτρα για την ενίσχυση των, του κώδικα σύνορων Σέγγεν, την οδηγία για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, το σύστημα εισόδου-εξόδου και την προπτική ε, ε, προοπτική του ATS. Νομίζω ότι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά ως αντίλογο ε, σε αυτούς που ε, με λαϊκισμό ή με προπαγάνδα προωθούν τα όσα κάνει το Ισλαμικό κράτος. Επίσης να πω ότι συμφωνώ απολύτως με την κυρία Σαρτζεντίνη που λέει ότι δεν ε, αρκεί απλώς να ασφαλίσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Αυτό δεν μπορεί να είναι το τέλος στα όσα προσπαθούμε να κάνουμε. Ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την προσαρμοστικότητα της κοινωνίας μας ε, και τις προκλήσεις που υπάρχουν για ριζοσπαστικοποίηση ε, σε κάθε χώρα και πώς μπορούμε να πατάξουμε αυτή τη ριζοσπαστικοποίηση. αναφέρομαι συστηματικά σε αυτό και θα συνεχίσω να αναφέρομαι γιατί για μένα αποτελεί το επίκεντρο των προσπαθειών μας. Αύριο Υπάρχει μια διάσκεψη την οποία φιλοξενεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα συζητήσει τις αποτελεσματικές ε, δομές ε, ε, και μορφές παρέμβασης. Σας το ανέφερα προηγουμένως. Είναι οργανωμένη προσέγγιση για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και θα ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να συστήσουν και να υποστηρίξουν ένα αποθετήριο βέλτιστων πρακτικών ώστε να μπορέσουμε να βρούμε και την κοινωνία των πολιτών και ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην πηγή του προβλήματος, να δούμε τι διδάγματα μπορούμε να αντιλήσουμε από αυτούς και να υπάρχει και ένα εθνικό σημείο επαφής, ώστε κάποιος, ένα άλλο κράτος μέλος που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, να ξέρει πού να στραφεί, προκειμένου να λάβει βοήθεια και συμβουλές από ανθρώπους ισότιμους με αυτόν και υπάρχει και μια νέα πρωτοβουλία που λέγεται Run Young προκειμένου να ενθαρρύνουμε και να ενδυναμώσουμε τους νέους ανθρώπους για να ε, αναλάβουν πιο δραστήριο ρόλο για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Διότι ε, το συζητήσαμε και στο παρελθόν, έχετε εργαστεί από αυτού ότι πρέπει να υπάρχει και δέσμευση μέσω της παιδείας και μέσω άλλων μέσων για τα νέα παιδιά. Η πεποίθησή μου είναι ότι Κάποιοι από τους καλύτερους πρέσβεις για το έργο αυτό για τους νέους είναι οι ίδιοι οι νέοι και πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να συμμετέχουν πλήρως σε αυτό, πέραν των όσων πρέπει να κάνουμε για την ριζοσπαστικοποίηση αυτή καθεαυτή. Κάποιοι από εσά αναφέρθηκαν και στο PNR, στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών των επιβατών. Δεν θέλω ε, να σχολιάσω τις συζητήσεις που έγιναν όταν ε, διατυπώνατε άποψη για το ε, PNR. Το ξέρω ότι δεν είναι όλοι ε, θειασότες ε, της ε, αυτή. Πολλοί δεν πιστεύουν ότι είναι τέλεια τα όσα έχουν γίνει. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να κάνω ως επόμενο βήμα και ως πρώτο βήμα τελικά κατά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των όσων έχουν συμφωνηθεί είναι να εφαρμόσουμε αυτά που έχουν ε, συμφωνηθεί. Διότι πώς θα διαμορφώσουμε άποψη ε, για τα ε, στοιχεία, γιατί πολύ αναφερθήκατε στις αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει στοιχείων, εάν δεν δούμε τι γίνεται με την εφαρμογή του συστήματος. Επομένως, θα υπάρξει ένα σχέδιο εφαρμογής, διότι συμφωνώ κυρία Σίπελ και άλλοι ότι δεν αρκεί τα κράτη-μέλη ε, ε, καθυστερούν ε, στην εφαρμογή και μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα διανύμουμε μία έκθεση και σε εσά και στα κράτη-μέλη η οποία στόχο έχει να δώσει κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη-μέλη για τη μεταφορά της συγκεκριμένη οδηγίας θα περιλαμβάνει μία σειρά από ορόσημα και δράσεις που θεωρούμε ότι αποτελούν τα βασικά στοιχεία για τη σύσταση του συστήματος PANR και ε, τη συμμόρφωση με την οδηγία. Παραδείγματο χάρη, πρέπει να υπάρχει η λεγόμενη PAU. Πρέπει να υπάρχει μία αρχή η οποία θα είναι η αρμόδια PAU στη η χώρα σας, ε, πού θα είναι, πώς θα λειτουργεί. Πρέπει επίσης να υπάρξει μια τεχνική λύση για την επεξεργασία των στοιχείων PNR. Ε, να στελεχωθεί η PIU και ε, να διοριστεί και υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Πρέπει να βρείτε ποια θα είναι η αρμόδια αρχή η οποία θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει δεδομένα PNR. Πρέπει επίσης να λάβετε ε, μέτρα ώστε να υπάρχουν σύνδεσμοι με ε, αεροπορικές εταιρείες ώστε να λαμβάνετε τις πληροφορίες και φυσικά ε, με τρόπο και μορφή που θα μπορείτε να τα επεξεργαστείτε και από εκεί και πέρα να τα μοιραστείτε και με άλλους. Και όλα αυτά φυσικά απαιτούν και πρακτικά μέτρα και σε πολλές περιπτώσεις και μέτρα σε εθνική νομοθεσία. Αυτά βέβαια δεν πρέπει απαραίτητα να γίνουν με χρονολογική σειρά ε, οι βαθμιδών, αλλά πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να αντιμετωπίσετε όλα αυτά τα ζητήματα εάν θέλετε να προχωρήσετε με την εφαρμογή. Και θέλουμε να δούμε πού βρίσκονται τα κράτη-μέλη, πού θα πρέπει να γίνει περαιτέρω προσπάθεια και τι μπορούμε να κάνουμε εμεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά έργανα για να βοηθήσουν. Με τα χαρά να τα συζητήσω αυτά μαζί σας. Τώρα, για τα ευρύτερα ζητήματα αξιολόγηση τη αποτελεσματικότητα, Δεν μπορώ να πάω το χρόνο πίσω. Δεν θα σταματήσω όμως και το χρόνο, γιατί δεν νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια αποτελεσματική διαδικασία για να υπάρχουν κάποια διδάγματα και στο μέτρο του δυνατού να διαμορφώνουμε και μια άποψη βάση ε, στοιχείων. Γι' αυτό ακριβώς και θα στήσω μια δομή για την αξιολόγηση αυτή και θα ήθελα να ε, γίνει αυτό με τη βοήθειά σας. Θα υπάρξουν ε, κάποιες ιδέες για κάποια θεματικά εργαστήρια νομίζω, για να δούμε ε, ποιες είναι οι θεματικές ενότητες που μας αφορούν και τι θέματα πρέπει να εξετάσουμε και αν έχετε κάποιες προτάσεις για το πώς μπορούμε να τα διαρθρώσουμε όλα αυτά, ε, μπορούμε κάλλιστα να τις ακούσουμε και όταν θα ολοκληρωθούν αυτά τα εργαστήρια πιστεύω ότι πραγματικά θα υπάρχει συνεργασία μαζί σας. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε κάθε στοιχείο της αξιολόγησης. Είμαι βέβαιος ότι θα κάνετε κριτική αξιολόγηση της αξιολόγησης του χρόνου, αλλά σας ε, προτρέπω να συμμετέχετε στην όλη διαδικασία της ε, αξιολόγησης και ελπίζω θα ε, βοηθήσει και για σημεία βελτίωσης. Ε, προσωπικά εγώ δεν έχω ιδεολογικό πρόβλημα να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι σε κάποιους τομείς ε, δεν χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα, μπορεί να κάνουμε και λιγότερα. Δεν έχω και ιδεολογικό θέμα να πω ότι κάποια πράγματα που γίνονται ίσως πρέπει να σταματήσουν ή πρέπει να γίνουν με άλλο τρόπο ή πρέπει να αλλάξουν. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Όσον αφορά τα πυροβόλα όπλα, το θέμα που ανέφερε κάποιος ε, εκ των βουλευτών, Ζητώ συγγνώμη, εγώ έχω ενθουσιώδη άποψη για τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι θα σας εξέπλητε άλλοτε, ε, άλλωστε να μην υποστηρίξω τη θέση της Επιτροπής. Αλλά όπως ε, σας είπα, Πραγματικά θέλω πλέον να βρούμε έναν τρόπο να συμφωνήσουμε μαζί για το τι ακριβώς θα κάνουμε στον τομέα αυτό, διότι πιστεύω ότι σύντομα, ένα χρόνο μετά και από τα γεγονότα στον Πατακλάν, θα είναι ακόμα δύσκολο να εξηγήσουμε δημοσίως γιατί σταματήσαμε προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία, θα πρέπει να είναι μια συμφωνία στην οποία ε, θα μπορούν όλες οι πλευρές να πούν ότι ε, την υποστηρίζουν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θέλω εγώ να υπονομεύσω την πολύ αναλυτική συζήτηση που γίνεται για το πώς μπορούμε να εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους. Ελπίζω όμως να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία σύντομα και ότι η συμφωνία αυτή θα περιορίσει την κυκλοφορία των πλήρως αυτόματων και ε, των ε, ε, ημιοαυτόματων όπλων κατόπιν μετατροπής και να μπορεί να επιτρέπεται μόνο η νόμιμη χρήση τους σε διάφορα σημεία. Αυτή νομίζω ότι είναι η φιλοδοξία μας και ε, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν 11 συνάδελφοι που είχαν ζητήσει τον λόγο. Είναι αδύνατον. Και δεν μπορώ να προσθέσω άλλους. Θα ήθελα να ζητήσω να ε, μη μακρηγορήσετε έτσι ώστε να ακούσουμε όλους. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ ε, κύριε Επιτροπέ για την παρουσία σας εδώ και πράγματι χαίρομαι που ε, θα αντιμετωπίσετε και το ζήτημα των τοξιδιωτικών αγράφων. Είναι ένα σημαντικό θέμα για το οποίο δεν έχουμε ε, επαρκείς αρμοδιότητες. Το ζήτημα της Ένωσης για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας είναι ένα ζήτημα στο οποίο θα πρέπει να δούμε τι έχουμε πετύχει και πώς θα βελτιωθούμε. Το σύστημα SIS-2 είναι κατά την άποψή μου το καλύτερο δυνατόν παράδειγμα. Γιατί είναι, κεντρικό και αποτελεσματικό, επομένως θα έπρεπε να βελτιωθεί για να ε, βελτιωθεί και η ασφάλεια του επίπεδου ασφάλειας που παρέχουμε στους Ευρωπαίους πολίτες. Σύντομα θα έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει και στοιχεία ε, δακτυλοσκοπικά. Ωστόσο, προβλέπεται η υποχρέωση των κρατών μελών να εισάγουν στο σύστημα alert, ειδοποίησης. Θα ήθελα γι' αυτό το λόγο να σας ρωτήσω ποιες τεχνικές βελτιώσεις προβλέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο SIS2. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Τσενίτση, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Κίνγκ για την παρουσία του εδώ σήμερα. Πρέπει να πω ότι μου άρεσε η παρέμβασή του, γιατί είμαι και σκιώδη εισηγήτρια των σοσιαλιστών ε, ε, για την οδηγία για την τρομοκρατία. Χαίρομαι που αρχίσατε να συζητάτε την οδηγία και είπατε ότι θέλετε το συντομότερο δυνατόν να καθορίσουμε το κείμενο τη οδηγία. και εγώ είμαι βέβαιη ότι θα υπάρχει ένα σφαιρικό πλαίσιο στο ποινικό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την τρομοκρατία. Χαίρομαι που ξεκινήσατε αναφέροντα ε, τη στήριξη προς τα θύματα, διότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Αλλά Επίσης, ε, θεωρώ ότι αυτό το πλαίσιο ποινικού δικαίου θα πρέπει να υποστηρίζεται και από μια μακροχρόνια στρατηγική πρόληψης. Αναφερθήκατε στην πρόληψη κυρίως ως μορφή εκπαίδευσης των νέων. Υπάρχει όμως και ένα πρόβλημα ριζοσπαστικοποίησης εντός των φυλακών. Επομένως θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσον στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο και επ' αυτού. Μια άλλη πτυχή και χαίρομαι που την αναφέρατε είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και η περαιτέρω στήριξη που θέλουμε να δώσουμε προς τις διάφορες υπηρεσίες Eurojust, ε, Europol και η Ιουλίζα, την οποία επισκέφθηκα την προηγούμενη εβδομάδα και εκτίμησα ιδιαίτερο τη δυνατότητα εφαρμογής και ε, υλοποίηση τη δραστηριότητά τη. Όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών όμω, ρεαλιστικά αντικειμενικά υπάρχει κάποια αντίσταση από πλευράς ε, κάποιων χωρών για την ανταλλαγή πληροφοριών. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν πέραν της εφαρμογής ε, και της ε, βοήθειας προς τις υπηρεσίες. Ε, και κάτι ακόμα πολύ γρήγορα, μια πτυχή που εκτιμώ ιδιαίτερα είναι η αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία βεβαίως και αυτή πρέπει να συμπεριληφθεί στην οδηγία για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και για να ολοκληρώσω και ολοκληρώνω αμέσω. θα ήθελα να σας ρωτήσω και το εξής. Αναφερθήκατε στου ξένου μαχητέ. Θεωρείτε ότι πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες σε θέματα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και με ποιες χώρες ε, πιθανόν θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόνι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε, για αυτή την πλήρη παρουσίαση που κάλεψε όλα τα θέματα της Ένωσης, της ασφάλειας στην Ένωση. Ακούστηκαν πολλά ερωτήματα. Ε, εγώ θα το θέσω ανοιχτά. Ποια είναι τα εμπόδια που διαπιστώνετε. Τι περιμένετε από τα κράτη-μέλη. Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν προβλήματα στο επίπεδο των κρατών μελών όταν ε, ξεκινάει η εφαρμογή των οδηγιών, όταν αρχίζουμε να συζητάμε για την ανταλλαγή πληροφοριών ή δεδομένων. Εκεί ξεκινάνε να υπάρχουν προβλήματα. Χρειάζεται λοιπόν να γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματα αυτά, όχι για να έχουμε κάποια κράτη-μέλη που θα είναι δακτυλοδεικτούμενα, αλλά για να έχουμε τη δυνατότητα ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ασκήσουμε πίεση στις εθνικές κυβερνήσεις. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Εντφέλτ. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επιτροπή για την παρουσία σας εδώ. Με χαροποιεί το γεγονό ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στη συνεργασία σα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαίρομαι που έχετε, ε, έχετε παρευρεθεί σε επιτροπή του Κοινοβουλίου περισσότερε φορέ από ορισμένου συναδέλφου σα που έχουν αναλάβει τα καθήκοντά του εδώ και δύο χρόνια, να το πούμε αυτό. Χαίρομαι επίση για το γεγονό ότι ε, ακολουθείτε την σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το ψήφισμα του 2011 ότι χρειάζεται δηλαδή να γίνει μια γενική και συνολική αξιολόγηση της πολιτικής μας για την ασφάλεια. Και αν σας ενδιαφέρει ευχαρίστω να συνεισφέρω και εγώ σε αυτή την αξιολόγηση με τις προτάσεις μας. Τώρα, μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση για το PNR. 130 εκατομμύρια ευρώ έχουν δαπανηθεί από, τους, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σύστημα PNR συνολικότερα. Τα 10 εκατομμύρια από αυτά Η ομιλήτρια διαπίστωσε ότι κάπου υπάρχει ένα ενδιαφέρον βίντεο. 10 λοιπόν εκατομμύρια ευρώ είχαν προβλεφθεί να δαπανηθούν για τη διασύνδεση εθνικών συστημάτων. Θα ήθελα να έχω περισσότερες ε, πληροφορίες περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο δαπανήθηκαν τα χρήματα αυτά, για την συγχρηματοδότηση από την πλευρά των κρατών μελών, ιδιαίτερα στο ζήτημα της διαλειτουργικότητας. Δεν χρειάζεται να μου δώσετε τώρα τα στοιχεία, μπορεί και γραπτό αργότερα. Και ε, ε, ε ποια ήταν η πολιτική, γιατί. Ε, τα κράτη-μέλη είχαν αρχίσει να συλλέγουν δεδομένα ήδη από την πρώτη ημέρα και δεν είχαν ε, παρουσιάσει στοιχεία όπως τα όφυλαν σε συμφωνία με τις πολιτικές μας για τη διατήρηση δεδομένων. Ε, και το ερώτημα που σας θέτω είναι το εξή. Από πλευράς ασφαλείας, δεν πιστεύετε ότι είναι μεγάλος κίνδυνος να έχουμε κάποια κράτη-μέλη τα οποία υπονομεύουν το κράτος δικαίου. Με άλλα λόγια, πώς ζητάμε και πώς περιμένουμε από τα κράτη-μέλη να εμπιστεύονται το ένα από το άλλο όταν η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει να εξετάζει την πιθανότητα να κινήσει τις διαδικασίες για την παραβίαση του κράτους δικαίου σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος. και θα κλείσω κύριε Πρόεδρε, έχουμε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έχουν δαπανηθεί για την καταπολέμηση της τροποκρατίας. Σε ορισμένες χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία έχουν ξεκινήσει ε, έρευνες α, Διακινούνται λοιπόν τεράστια χρηματικά ποσά. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και κάποιες χώρες όπως η Ολλανδία που ίσως να είναι κέντρο τρομοκρατίας και εγώ πραγματικά είχα εκπλαγεί όταν διάφασα τις σχετικά δημοσιεύματα. Ε, λοιπόν, διακινούνται τόσο μεγάλα με χρηματικά ε, ποσά. Θα ήθελα να ε, μου ενημερώσετε αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να ε, επευθυνθεί και να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη που έχουν ξεκινήσει τέτοιες έρευνες. Ο Ντάλτον. Εμείς είχαμε υποστηρίξει την πρόταση της Επιτροπής για το PNR και θα θέλαμε να σας ενθαρρύνουμε, να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέσει τα κρατημέλη που δεν το έχουν κάνει ακόμα να προχωρήσουν στην εφαρμογή του συστήματος. Τώρα, όσον αφορά την ρίζοσπαστικοποίηση, χαίρομαι που ακούω που συζητάμε για την ε, ε, ε απεύθυνση στους ε, νέους ε, στη βάση. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και το ζήτημα του αθλητισμού. Γιατί εκεί έχουμε μια ευκαιρία να απευθυνθούμε σε ανθρώπους οι οποίοι δυνητικά θα μπορούσαν να ριζοσπαστικοποιηθούν, να ε, συνεργαστούμε με τις ε, ε, αθλητικές ομάδες, τις επαγγελματικές αθλητικές ομάδες. Επίσης, φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό η ριζοσπαστικοποίηση ε, γίνεται στις φυλακές. Αυτό το διαπιστώνουμε σε διάφορα κράτη-μέλη, το οποίο βέβαια σχετίζεται και με τις συνθήκες κράτησης. Θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό και τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα. Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας φυσικά δεν μπορεί παρά να είναι κατά κύριο λόγο ε, αμυντικού χαρακτήρα, αλλά υπάρχουν και κάποιες κινήσεις ε, πρόληψης, αν θέλετε, και θα ήθελα να με ενημερώσετε από αυτού τι είδους ε, συνεργασίες σκοπεύετε να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε με τρίτες χώρες ανά τον κόσμο για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Κύριε Γκάλ, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Όλοι συμφωνούμε ότι το χαρτοφυλάκιο σας είναι ιδιαίτερα σημαντικό ιδιαίτερα στην σημερινή ε, χρονική συγκυρία. Εγώ θα ήθελα να σα ρωτήσω κάτι για την έκθεση τη ομάδα επιγνωμένων υψηλού επίπεδου για τη διαλειτουργικότητα και τα πληροφοριακά συστήματα. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα επόμενα βήματα μετά την έκθεση αυτή. Θα κάνετε κάποιο σχέδιο εφαρμογή μέτρων ή μήπω σκοπεύετε να αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία. Για το PNR, το ερώτημά μου εμένα είναι σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, σε ποιο σημείο εφαρμογής. και για την ζήτημα της ριζοσπαστικοποίησης, το οποίο όλοι συμφωνούμε είναι πάρα πολύ σημαντικό, πώς σκοπεύετε να κατεπολεμήσετε τη ριζοσπαστικοποίηση στο ίντερνετ. Ευχαριστούμε. Ε, κύριε Γκρίνσπεκ, εγώ θα είμαι σύντομη. Στην ακρόασή σας πριν από δύο μήνες είχαμε συζητήσει για το ζήτημα της ασφάλειας στο διαδίκτυο, της κυβερνοασφάλειας. Και είχατε αναφέρει μια έννοια η οποία μου είχε φανεί κάπως ιδιαίτερη, κάπως περίεργη, το ζήτημα της ανθεκτικότητας της, ε, στην, στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Θα ήθελα να ε, λίγο, να μας δώσετε λίγες περισσότερες πληροφορίες από αυτού, τι σκοπεύετε να κάνετε στον τομέα για την αντιμετώπιση του hacking, για την αντιμετώπιση της υποκλοπής δεδομένων, ε, της επιθέσεις, ε, της κυβερνοεπιθέσεις. Δεν είμαι ειδική στον τομέα, είναι, ε, κάπως να παρακολουθώ αυτές τις ε, συζητήσεις, αλλά με έχει ιδιαίτερα ε, δημιουργήσει μια ανησυχία το ζήτημα της ε, χρήσης του ίντερνετ των προγμάτων ε, και της χρήσης ε, αυτής του οδού για την υλοποίηση τρομοκρατικών επιθέσεων. Ο κύριος Ντεπχέ. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τρία θέματα θέλω να θίξω. Πρώτον, είπατε ότι θα ενισχύσετε τις ε, προσπάθειές σας για να υλοποιηθεί το PNR. Βεβαίως, καιρός είναι, δέκα χρόνια το συζητάμε και ακόμα δεν είναι... Ε, δεν εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη. Έχουμε δύο που το χρησιμοποιούν, δύο, τρία, ε, μέχρι το τέλος της χρονιάς. Σύμφωνα με το έγγραφο το ενημερωτικό που διάβασα, τρεις θα χρησιμοποιούν το σύστημα, τρία κράτη-μέλη θα χρησιμοποιούν το σύστημα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτό είναι σκανδαλώδες κατά την άποψή μου. Δεύτερο θέμα. Είχα θέσει ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις, υπο, τις υποχρεώσεις ή τις ε, προϋποθέσεις μάλλον για την ανταλλαγή δεδομένων PNR. Η απάντηση που είχα λάβει είναι ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σκόπευε να δημιουργήσει ένα, μια λίστα τέτοιων κριτηρίων για την ανταλλαγή αυτών των ε, στοιχείων, γιατί αυτό θα περιόριζε το τη δυνατότητα των κρατομελών να αποφασίζουν ποια είναι τα δεδομένα τα οποία θέλουν να ανταλλάσσουν. Και πώς θα προχωρήσουμε έτσι όμως. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μια ανταλλαγή των δεδομένων που είναι τα δεδομένα που θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία. Αυτά δεν είναι τα δεδομένα που θα ήταν υποχρεωτικό και θα οφείλαμε όλοι να ανταλλάσσουμε. Ωραία. Για τους συστηματικούς έλεγχους στο χώρο Σέγγεν ακόμα και για τους υπο, ε, υπηκόους της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Έχουμε 27 διαφορετικά συστήματα ταξιδιωτικών εγγράφων, ταξι, ε, ταυτοτήτων, ε, ταυτοποίησης των ανθρώπων. Μιλάω για 27 κρατημέλη για να μην μιλήσω και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι 27 διαφορετικά. Δεν θα μπορούσαμε κάπως να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Γνωρίζουμε ότι οι ταυτότητες είναι το ταξιδιωτικό έγγραφο, το έγγραφο ε, το οποίο πλαστογραφείται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Δεν θα έπρεπε κάπως να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα υπό το πρίσμα της ενίσχυσης της ασφαλείας μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λόριστον. Σα ευχαριστώ πολύ που μας δώσατε τις πληροφορίες αυτές και η ερώτησή μου συνδέεται με την ερώτηση της κυρίας Κρίσπεκ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τι νέε εξελίξει, διότι ε, βλέπουμε τις γρήγορε εξελίξεις του ίντερνετ των πραγμάτων, ε, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις ταχυδρομικέ υπηρεσίε στον ιδιωτικό τομέα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε γενικότερα την ψηφιακή ασφάλεια. Υπάρχουν νέες εξελίξεις. Συνεργάζεστε με τον Επίτροπο Επιψηφιακών Θεμάτων για το θέμα αυτό, διότι βλέπουμε νέες απειλές. Και η δεύτερη μου ερώτηση έχει να κάνει με την καταπολέμηση της ε, ριζοσπαστικοποίησης. Ε, πρόκειται για έναν ε, πόλεμο πληροφοριών από τρίτες χώρες. Δεν συνδέεται με την αντικατασκοπία, συνδέεται με... Πρέπει να κοιτάξουμε τις άμεσες ενέργειες και Πρέπει να οικοδομήσουμε δυναμικό, να είμαστε ανθεκτικοί. Λάβαμε από την Europol πληροφορίες σχετικά με την ε, το, το νέο τμήμα ε, που ασχολείται ακριβώς με αυτόν ε, τον πόλεμο πληροφοριών. Μήπως μπορείτε να αναφερθείτε σε αυτό και την διεθνή πτυχή του θέματος αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Στιέστεμερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο. Η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα στον αγώνα κατά εκείνων που ε, επιχειρούν κατά τις ελευθερίες μας. Αλλά η ελευθερία είναι ε, το αντίδοτο στην τρομοκρατία. Θα σας πω κάτι που σίγουρα δεν θα θέλετε να το ακούσετε. Η Μουσούλη είναι επερκυκλωμένοι, ε, η ράκα αποτελεί αντικείμενο επίθεσης και ε, αρχίζουν να βραχικοκλώνονται οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ Ιράκας και Μοσούλης. Ε, η δράση του Ισλαμικού κράτους σίγουρα θα τους οδηγήσει σε μία αντίδραση χωρίς καμία διάκριση, αυξημένη και βίαιη στην περιοχή μας ως τρόπος για να αντισταθμίσουν την απώλεια και να ε, δημιουργήσουν ψευδεστήσει ψευδεστήσεις σε αυτούς που είναι ήδη παραστρατημένοι και ζουν σε έναν διαφορετικό κόσμο. Ξέρω λοιπόν που βρίσκονται οι ακαδημαϊκές συζητήσεις και οι συζητήσεις στα κοινοβούλια και ε, εδώ να πω ότι ναι μεν επικροτώ τις προσπάθειές μας θα ήθελα ε, να σταθώ όμως σε κάποιες ε, πτυχές για αυτές τις κοινέ προσπάθειες. Καταρχάς να πω ότι συμφωνώ με την κυρία Σαρχεντίνη. Δεν μπορούμε μόνο να δεσμεύσουμε, ε, να, να, να συνδυάσουμε συγγνώμη, τη σχέση τρομοκρατίας και ξεπλήματος χρήματος, δεν έχουμε και κανένα μέσο για να εξουδετερώσουμε αυτή τη σχέση. Και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε τίποτα. Ε, κύριε Επίτροπε, λοιπόν, θα ήθελα να ξέρω αυτό που είπατε εσείς ότι θα περιπλέξετε τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, πώς θα το επιτύχετε. Ο, τέλος, όσον αφορά το θέμα εισόδου-εξόδου, αρκετό καιρό ασχολούμαι με τα σημεία εισόδου-εξόδου και είπατε εσείς ότι σύντομα θα μας παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σύστημα έγκρισης ταξιδίων. Θα ήθελα να ξέρω τι ακριβώς ε, θα περιλαμβάνει αυτό το σύστημα. Επίσης να πω ότι αντιλαμβάνομαι πολύ καλά τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ ε, μιας ταυτότητας και ενός ταξιδιωτικού εγγράφου. Αυτό το οποίο πρέπει να βελτιώσουμε είναι τα ταξιδιωτικά έγγραφα μέσω ε, μιας ε, ε, κοινοτικής ε, κρυπτογράφησης, κωδικοποίησης. Θα μπορούσα να συνεχίσω να τα συζητώ τα θέματα, αλλά νομίζω ότι χρειάζομαι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις. Η κυρία Γκαμπριέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε, σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας και ε, σας ευχαριστώ και για τις ε, πολύ ε, επίκαιρες πληροφορίες που μας δίνετε. Δύο πράγματα όσον αφορά την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Νομίζω ότι πολύ σωστά είπατε, έγινε πολύ σημαντική δουλειά και πρέπει... Ε, το δίκτυο ΟΡΑΝ να το εκμεταλλευτούν τα κράτη-μέλη. Επίσης, πρέπει να δραστηριοποιηθούμε σε το τοπικό επίπεδο. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι οι δήμαρχοι, οι τοπικές αρχές μπορούν να συνεισφέρουν και θα ήθελα να ξέρω τι θέλετε να κάνετε σε αυτό το επίπεδο, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι δράσεις που κάνουμε είναι στο ύψο των προκλήσεων. Μία ερώτηση όσον αφορά την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στο διαδίκτυο οι δράσεις της Interpol μέσω διαδικτύου φαίνονται ε, αποτελεσματικές. Πώς μπορείτε εσείς να πείσετε τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν περισσότερο σε αυτές τις δράσεις. Επίσης, ε, πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν και στο θέμα αυτό, αλλά με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η διαλειτουργικότητα των δεδομένων και η συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών ε, είμαι υπέρ της ε, σύστασης της ομάδας εμπειρογνωμόνων, αλλά θα ήθελα να ξέρω ποιο είναι το δέλεαρ και ποια είναι η τιμωρία για να αναλάβουν τις ευθύνε του στα κράτη-μέλη. Και επίσης θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται με τη δυνατότητα επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων. Είναι άχρηστο να έχουμε περισσότερα δεδομένα, αν δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσετε. Έχετε μια αξιολόγηση για τις ελλείψεις ή τα προβλήματα που υπάρχουν για τα μέσα ή τα εργαλεία που χρειαζόμαστε σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ. Thank you. And, um, Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χιμένεθ Βεθερίλ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και θεωρώ ότι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας είναι πολύ σημαντική για να προβάλλουμε ε, την αύξηση της ασφάλειας ενώπιον και αυτής της απειλής της τρομοκρατίας που αντιμετωπίζουμε. Ε, ορισμένες φορές δεν θέλουμε να τα ακούσουμε γιατί είναι πολύ σκληρό και κανείς δεν θέλει να νιώσει ότι απειλείται. Εγώ μόλις έρθα από τα Ηνωμένα Έθνη και ήμουνα και με τον ε, ε επικεφαλής ε, της ε, Task Force για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και μου έλεγε ότι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα είναι το Ισλαμικό κράτος. Όταν θα φύγουν από τη Μοσούλη πώς θα δραστηριοποιηθούν στην Ευρώπη. Δεν είναι τίποτα γενοφανές αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να δράσουμε. Δεν υπάρχει ορισμός της τρομοκρατίας. Δεν υπάρχει ε, ενότητα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας ούτε εδώ στην Ευρώπη, πολλό δε μάλλον όταν πρέπει να συνεργαστούμε με τα Ηνωμένα Έθνη ή με άλλους διεθνείς οργανισμούς, γιατί δεν υπάρχει ένας κοινό ορισμός της τρομοκρατίας. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να γίνουν τέσσερα πράγματα. Πρόληψη, προστασία, συνέχεια και απάντηση. Και πρέπει να γίνουν με αυτή τη σειρά. Και όχι μόνο εδώ, αλλά πρέπει να γίνει και όπως σας είπα και με τα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να καταφέρουμε κάτι και με τρίτες χώρες. Επίσης, θα ήθελα να πω επιτέλους, ε, διότι δεν έχω αρκετό χρόνο, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα θύματα να γίνει κάτι. Ε, υπάρχει μια οδηγία αυτή τη στιγμή, στην οποία θα έχουν μεγάλη σημασία τα θύματα της τρομοκρατίας μεν, αλλά δεν υπάρχει ορισμός για το θύμα. Δεν θέλησε κανείς να συμπεριλάβει ορισμό στο κείμενο. Ε, στις περισσότερες τροπολογίες ε, που κατέθεσα εγώ ε, δεν έγιναν αποδεκτές. Πρέπει να επιμένουμε για τη σημασία των θυμάτων δεν είναι μόνο θέμα αλληλεγγύης, είναι θέμα και το γεγονότος ότι είναι ενεργά στοιχεία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το κέντρο συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη στήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας, γιατί όταν υπάρχει μια επίθεση σε μια χώρα είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει κεντρικό συντονισμός. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Θα σας παρακαλούσα να προσπαθήσετε να απαντήσετε σε ερωτήσεις αυτές. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Ξέρω ότι σε πολλές ε, από τις ερωτήσεις αυτές μπορείτε να απαντήσετε γραπτώς. Θα σας παρακαλούσα όμως να προσπαθήσετε να καλύψετε όσο γίνεται περισσότερες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και πάλι για το ενδιαφέρον σας ε, για τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι ένα από τα ωφέλη αυτών των ε, διαλόγων ε, είναι ότι ανακαλύπτω πράγματα και ελπίζω να ε, συνεχιστούν σε τακτική βάση οι διάλογοι αυτοί. όσον αφορά διάφορα θέματα που αναφέρθηκαν, και συγχωρήστε με αν ε, δεν καταφέρω να συνδέσω το κάθε θέμα με το σωστό όνομα λόγω ε, της πίεσης του χρόνου από πλευράς του Προέδρου. 11 και 45 έχουμε ψηφοφορία. Αν συμφωνείτε μπορούμε να ξεπεράσουμε λίγο το χρόνο. Καταρχάς ε, έχουμε μια σειρά ερωτήσεων που συνδέονται με τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Πολλοί έθεσαν ε, σχετική ερώτηση και αναφέρθηκαν και διάφορες πτυχές του θέματος αυτού. Θα ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι είναι πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιοι ε, περιορισμοί όσον αφορά τις αρμοδιότητες που θα πρέπει να σεβαστούμε στον τομέα αυτόν όπως και σε όλους τους τομείς. Υπάρχουν όμως και θέματα ασφαλείας. Ε, τα στα οποία θα ήθελα να σημειώσουμε πρόοδο σε συνεργασία με την συναδελφό μου την κυρία Γιούροβα. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν με το δελτίο ταυτότητάς τους να ε, ταξιδέψουν ε, εντός της ε, περιοχής Σέγγεν καθώς και σε κάποιες τρίτες χώρες. Και πώς να το θέσω ευγενικά. Δεν πληρούν ε, όλες οι εθνικές ταυτότητες ε, τις ίδιες προϋποθέσεις ασφαλείας. Κάποιες είναι πιο εύκολο να πλαστογραφηθούν από άλλες. Και αυτό δεν είναι μόνο εθνικό πρόβλημα. Και νομίζω ότι κάτι θα πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να συμφωνήσω με την ε, συναδελφό μου την Επιτροπό Γιουρόβα στην ε, μελέτη αντικτύπου που ε, θέλει να διενεργήσει πάνω στις ταυτότητες με στόχο πιθανές προτάσεις του χρόνου, το 2017. Διότι νομίζω ότι αυτό είναι θέμα ασφαλείας που ξεπερνάει τα σύνορα της κάθε χώρας και με αυτό συνδέονται και άλλα θέματα όπως είναι τα breeder documents τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε στο πλαίσιο αυτό. Τα, ε, πρόκειται για τα έγγραφα ε, με βάση τα οποία εκδίδονται άλλα επίσημα έγγραφα. Και επίσης, ε, ρωτήθηκε τι θα κάνουμε για το SIS. Έχουμε κάνει μια αξιολόγηση. με βάση την οποία θα προτείνουμε μια πρώτη σειρά τροπολογιών ε, για το σύστημα αυτό. Και λέω μια πρώτη σειρά, διότι νομίζω ότι θα υπάρξει η δεύτερη σειρά προτάσεων μετά από συζητήσεις μαζί σας. Ε, μετά τα, αφού ακούσουμε τα αποτελέσματα της ε, ε, ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου, αλλά θα συμπεριλάβουμε προτάσεις ε, για να μπορούμε να εντοπίζουμε ανθρώπους με βάση μόνο τα δαχτυλοσκοπικά ε, τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Επίσης, ένα νέο ε, σύστημα καταχώρησης για αγνώστου καταζητούμενου σε περίπτωση λέει, που έχουμε μόνο τα δαχτυλικά αποτυπώματα χωρίς όμως άλλα δεδομένα. Νομίζω ότι αυτό θα είναι χρήσιμο για την αντιμετώπιση του εγκλήματος και πιθανότατα και της τρομοκρατίας. Και φυσικά θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν οι διαδικασίες και ε, τα συστήματα ώστε ε, οι διαδικασίες αυτές ε, να μην κρατάνε περισσότερο από ότι είναι απολύτως απαραίτητο. Επίσης, μία δεύτερη σειρά προτάσεων για καλύτερη εφαρμογή ε, των αποφάσεων περί επιστροφής, ε, ζητώντας δηλαδή από τα κράτη-μέλη να εισάγουν τα απαραίτητα στοιχεία στο σύστημα, ώστε ε, αν έχει επιστραφεί κανείς ή αν έχει απαγόρευση εισόδου, αυτό να καταχωρίζεται, ώστε να μην μπορούν να επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει πάλι να φροντίσουμε τα προσωπικά δεδομένα να διατηρούνται μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν όμως κάποια συγκεκριμένα πράγματα που νομίζω μπορούμε να κάνουμε τώρα κατά την πρώτη αναθεώρηση του συστήματος ε, ΣΥΣ και πιθανότατα θα έχουμε μια δεύτερη σειρά προτάσεων του χρόνου. Επίσης, ε, κάποιοι ευρωβουλευτές και τελευταία η κυρία Χιμένε αναφέρθηκε στα θύματα, κάτι στο οποίο αναφέρθηκα και εγώ σύντομα στην αρχή της ε, παρεμβασή μου. Έχω συνομιλήσει με δίκτυο υποστήριξη των θυμάτων που νομίζω ότι κάνει εξαιρετική δουλειά και έχω δεσμευτεί να συνεργαστώ στενά μαζί τους, ε, να ε, συμμετάσχω και σε κάποιε από τι συναντήσεις του, ώστε να φροντίσουμε να διατηρήσουμε τα θύματα στο επίκεντρο κατά την ανάπτυξη αυτού του θεματολογίου. Υπάρχει όμως ένα συγκεκριμένο θέμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ. Πρόκειται για τη συνεργασία με τα θύματα για να ε, έχουμε αφηγήματα κατά της ριζοσπαστικοποίησης, διότι νομίζω ότι από τις πιο ισχυρές μαρτυρίες ε, που μπορούν ε, να μας βοηθήσουν στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης ε, προέρχονται από τα θύματα και το εννοώ αυτό με την ευρύτερη έννοια. Για παράδειγμα, οι μητέρες των παιδιών που έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί και έχουν πάει στην Συρία. Ο μόνος τρόπος όμως που μπορεί κανείς να συγκεντρώσει τέτοιες μαρτυρίες είναι όταν ε, ο ενδιαφερόμενος νιώθει ικανός να δώσει τη μαρτυρία αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να έχουμε μέτρα για να συνοδεύουμε τα, δίχτυα, τα θύματα της τρομοκρατίας μέχρι το σημείο που είναι διατεθειμένοι να εργαστούν για την ε, δημιουργία νέου αφηγήματος για την καταπολέμηση της ρίζοσπαστικοποίηση. και αυτό αποτελεί σημαντικό κομμάτι τη δουλειά μα για την καταπολέμηση της ρίζοσπαστικοποίηση. Όπω κάποιοι από εσά αναφέρατε, ζητήσατε περισσότερε λεπτομέρειε σχετικά με το τι θα κάνουμε στο πλαίσιο του ΡΑΝ. Για παράδειγμα, όσον αφορά τις φυλακές, τη χρήση του αθλητισμού, και θα προσέθετε και άλλα θέματα που συνδέονται με τις γυναίκες και τα παιδιά, διότι Εάν σημειωθεί πρόοδος, όπως όλοι ελπίζουμε, κατά του ΝΤΑΕΣ, ε, θα πρέπει να ε, σκεφτούμε όχι μόνο τους μαχητές ε, που θα επιστρέψουν, αλλά και οι οικογένειες που θα επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, τις οποίες πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε στο πλαίσιο του δικτύου κατά της ισοπαστικοποίησης. Επίσης, όσον αφορά τις φυλακές, ε, σε κάποια κράτη-μέλη ομαδοποιούνται οι κρατούμενοι, οι ριζοσπαστικοποιημένοι, ενώ σε άλλα κράτη-μέλη ε, μοιράζονται σε διαφορετικούς χώρους. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ανταλλαγή πρακτικών ε, στα θέματα αυτά και ιδιαίτερα με βάση τα κράτη-μέλη που έχουν κάνει την περισσότερη δουλειά στον τομέα αυτών. δεν έχουμε κάνει αρκετά όσον αφορά τη χρήση του αθλητισμού στις προσπάθειες μας κατά της ζωσπαστικοποίησης. Ε, όταν μιλάμε με ανθρώπους που το κάνουν αυτό στις διάφορες κοινότητες, λένε ακριβώς αυτό που είπατε και εσείς κύριε Ντόλτον. Ο ε, αθλητισμός είναι ένα από τους βασικούς τρόπους ε, να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους και ελπίζουμε ότι με αυτό το νέο δίκτυο του ΡΑΝ να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους και θα πρέπει να σκεφτούμε δημιουργικά σχετικά με την ε, χρήση του αθλητισμού και άλλες κοινωνικές δραστηριότητες ε, που ενώνουν τους ανθρώπους. Τέθηκαν διάφορες ερωτήσεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και το πώς θα χρησιμοποιήσουμε την ε, ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου και, και τι συνέχεια μπορούμε να δώσουμε στα, στα αποτελέσματα της ομάδας αυτής. Η πρώτη μου απάντηση είναι ότι θα επιταχύνουμε τι εργασίε, δηλαδή δεν θα περιμένουμε μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Θα έχουμε μια πρώτη έκθεση τώρα το Δεκέμβριο, την οποία θα συζητήσω μαζί σα και ε, αν υπάρχουν ε, πρακτικά στοιχεία της έκθεσης αυτής ε, στα οποία να μπορούμε να δώσουμε συνέχεια, όπως ανέφερα και νωρίτερα. Δεν θα περιμένουμε το επόμενο καλοκαίρι για να το κάνουμε αυτό. Θα εκπονήσουμε ένα πρόγραμμα για να προωθήσουμε τα ζητήματα αυτά σε συνεργασία μαζί σας τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με ριζοσπαστικοποίηση στο διαδίκτυο και θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της πρόκλησης αυτής και τη δουλειά που κάνουμε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τους ε, παρόχους υπηρεσιών του διαδικτύου στο πλαίσιο του ε, φόρουμ ε, του διαδικτύου του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, ενίσχυση των προσπαθειών μας κατά της ριζοσπαστικοποίησης ε, στο διαδίκτυο. Τον Δεκέμβριο έχουμε τη συνάντηση του φόρουμ και θα ήθελα να σας καλέσω να συμμετάσχετε εάν σας ε, ενδιαφέρει. Θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρό σας να ασχοληθεί με το θέμα αυτό, καθώς και με τις δραστηριότητες της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου. Πρόοδο ε, που έχουμε σημειώσει όσον αφορά το υλικό που δημοσιεύεται στο ίντερνετ ε, είναι καλή. Γνωρίζετε ε, το IU, τη Europol και τα πολλά στοιχεία που έχει εντοπίσει. Κάποια ο μέρος του υλικού είναι εγκληματικό, οπότε έπρεπε να αφαιρεθεί. Έχουμε ε, άλλες περιπτώσεις υλικού που δεν είναι ε, εγκληματικό, αλλά ε, με το οποίο πρέπει παρόλα αυτά να ασχοληθούμε. Και έχουμε ποσοστό επιτυχίας 90% και μπορεί το 50.000 να ακούγεται πολύ ωραίο νούμερο, παρόλα αυτά αποτελεί στο, σταγόνα στον ωκεανό σχετικά με τον όγκο του τέτοιου υλικού που υπάρχει στο διαδίκτυο. Ένα από τα πράγματα που ελπίζω ότι θα πετύχουμε μέσω του φόρουμ ε, του διαδικτύου είναι να διευρύνουμε το διάλογο με τους παρόχους υπηρεσιών ε, διαδικτύου ε, σχετικά με το υλικό αυτό και μάλιστα συμπεριλαμβανομένου υλικού που προέρχεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Λόριστα αναφέρθηκε στην συνεργασία με τρίτες χώρες και νομίζω ότι Υπάρχει σημαντική δουλειά που θα πρέπει να γίνει για να ε, διευρύνουμε τον διάλογό μας ε, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με τρίτες χώρες ε, για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε και την ριζοσπαστικοποίηση και την προπαγάνδα. Και συνομιλώ και με την Επίτροπο Μάλμστρομ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για να δούμε πώ μπορούμε να το πετύχουμε αυτό στου διαλόγου μα με τρίτε χώρε. Τέθηκαν κάποιε ερωτήσει σχετικά με τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία και στον προηγούμενο γύρο ερωτήσεων ε, δεν είχα... Ε, ε, δεν ήταν σκόπιμο που δεν απάντησα στην κυρία Σαρτζεντίνη. Υπάρχουν πράγματι κάποιες προκλήσεις για βελτίωση της δουλειάς μας στον τομέα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ακόμα και αν είναι σχετικά μικρά τα χρηματικά ποσά και ακόμα και αν οι τρόποι για την μεταφορά των χρημάτων αυτών είναι δύσκολο να ανοιχνευτούν, ασχολούμαστε με το θέμα και είχα συνομιλίες με την Europol σχετικά με την αποτελεσματικότητα ε, των ε, μηχανισμών τους όσον αφορά τον εντοπισμό το, της χρηματοδότησης ε, της τρομοκρατίας. Μάλιστα, Είμαι τόσο πεπισμένος σχετικά με ε, τις ε, δυνατές χρήσεις ε, της ανείχνευσης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που θα ήθελα πάρα πολύ να ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό, όχι σήμερα, αλλά κάποια άλλη στιγμή. Όσον αφορά την πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση σχετικά με τα εμπόδια που θα αντιμετωπίσουμε. Όσον αφορά τα εμπόδια που θα αντιμετωπίσουμε, τα γνωρίζετε, τα αναφέρατε στις διάφορες ερωτήσεις σας. Τα βασικά μας εμπόδια είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, ώστε να ξεπεραστεί η επιφύλαξη για τη συνεργασία, για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε τα συστήματα που τελικά θα μας επιτρέψει να έχουμε αποτελεσματική συνεργασία, είτε μιλάμε για το πλαίσιο του PNR, είτε για άλλα πλαίσια. Επίσης, ε, ο κύριος ε, Ντεπρέ ε, έδωσε πολύ σωστή ερώτηση. Δεν έχω την απάντηση αυτή τη στιγμή, θα το εξετάσουμε όμως. Και τρίτον, θέλουμε αποτελεσματική εφαρμογή των συστημάτων αυτών. Αυτές είναι οι προκλήσεις μας, δεν έχουν αλλάξει, τις γνωρίζουμε καλά και θα ήθελα πολύ σε συνεργασία μαζί σα να καταβάλουμε ε, ε, σωστή προσπάθεια για να τι αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε. Ε, ξεπεράσαμε λίγο το χρόνο δυστυχώ Να αναφέρω δύο πράγματα. Οι συνάδελφοι θα θυμούνται ότι θέλαμε να κάνουμε το διαρθρωμένο διάλογο για την ασφάλεια, που θέλω να το συζητήσω με τους συντονιστές βεβαίως, γιατί τα μέλη συζήτησαν θέματα με τον ε, για τα θέματα αυτά. Θα υπάρχει και συνέχεια και μας ενδιαφέρει και το θέμα των δεδομένων και της ασφάλειας. Σίγουρα χρειάζεται πιο διεξοδική συζήτηση από αυτού. Ε, δεν ε, ασχολούμαστε αποκλειστικά με αυτό. Πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα διαρθρωμένο διάλογο στον οποίο θα μπορούμε να εμβαθύνουμε περισσότερο στα θέματα αυτά. Θα τα συζητήσουμε με τους συντονιστές και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Νομίζω ότι για την πρώτη φορά ε, ε, πήγε πολύ καλά η παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μας δώσετε και ζητώ συγγνώμη από τους αδέλφους που δεν μπόρεσαν να θέσουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε. Συνάδελφοι, συγγνώμη για την καθυστέρηση για εκείνους που ήρθαν για τις ψηφοφορίες. Αν είστε έτοιμοι μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Να ελέγξω αν έχετε τις κάρτες σας. Αν δεν έχετε να μας το πείτε τώρα για να μπορέσουμε να ε, καταγράφουμε την ψήφο σας. Έχετε όλη την κάρτα σας, ωραία. Περνάμε στο σημείο 8 για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Συμβάσεις για την ε, προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου. Η κυρία Λόριστον είναι ε, η συγκήτρια. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι πριν από την ψηφοφορία. Πολύ σύντομα θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι είναι η πρώτη ευκαιρία για να συμμετέχουμε στην εφαρμογή της, του νέου κανονισμού για την προστασία δεδομένων. Και τρόπον την ε, θέτουμε το βηματισμό. Ο στόχος μας στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ήταν να καταφέρουμε ο κανονισμός για την προστασία δεδομένων να εφαρμοστεί πλήρως και να λαμβάνει υπόψη του όχι μόνο τη γενικότερη φράση με την επιφύλαξη, αλλά και τα προβλήματα που συμβαίνουν καθημερινά ε, κατά την ε, αντιμετώπιση ψηφιακού περιεχομένου για οτιδήποτε, από μουσική μέχρι λογισμικό. Σε όλες αυτές τις πρακτικές, ο κανονισμός για την προστασία δεδομένων θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο τμήμα τους. Ε, ευχαριστώ πολύ τους και συγητές, ε, την ομάδα. Υπήρχε μια θετική συνένεση και συγκατάθεση γιατί οι περισσότεροι συμμετείχαμε στη δημιουργία αυτού του κανονισμού και θεωρήσαμε ότι αποτελεί ευθύνη μας. Σας ευχαριστώ έλους. Ε, είναι περίπλοκο γιατί είναι καινούριο αυτό το στοιχείο αλλά ελπίζουμε ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ Μάριο. Περνάμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 88. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote isn't open. The vote is open now. Which is just enough time for Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, ίσα ίσα προλαβαίνει η Άννα Γκόμες να βάλει την κάρτα της. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 89. Τροπολογία 90, συγγνώμη. Άρχεται η ψηφοφορία. 90. Τροπολογία 90. 9-0. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 91. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 93. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όλα εντάξει. Συμβαστική τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Χαμογελώ, δεν ξέρω. Ε, χαίρεστε που δεν ψηφίζει ο κύριος Κοέγιο, εσείς το ΕΛΚ. Ε, εμείς διασκεδάζουμε με τον κύριο Κοέγιο, αλλά δεν ξέρω για τους υπόλοιπους. Συμβαστική τροπολογία 11, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Συμβαστική τροπολογία 11. Εγκρίνεται. Τροπολογία 106. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 112. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 113. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 115. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 116. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 117. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 122. Συγγνώμη. 121 και 122 είναι ταυτόσιμες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 123 και 124 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της προφορίας. Εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 128. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 131. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 132. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Α, πέραση της ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 134. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 135. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 136. Άρχεται η ψηφοφορία. Συγγνώμη. 136 και 137 μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 139. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 140. Υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία, συγγνώμη. Πέρας τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 141. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 142. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 151. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 152. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 153. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 154 και 155 ταυτόσημες άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 156 άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 157 άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση προφορίας. Απορρίπτεται. 158. Άρχεται η ψηφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 159. Άρχεται η ψηφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 160 και 161 ταυτόσημες, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της Εγκρίνεται. 162 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 172. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 173. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 174. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 175. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας της ψηφορίας. Εγκρίνεται. 176 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα έρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τι δούμε αν μπλοκ, επομένως ξεκινάμε. 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Closed. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 27. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 28. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Ε, κρίνεται. 29. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 30. Άρχεται η ψηφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 31. Άρχεται η ψηφορία. Πέραση τη ψηφοφορία, Απορρίπτεται. 32. Άρχεται η ψηφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 και 33 ταυτόσημες άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφορία. Εγκρίνεται. 34 άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 35 άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 36 άρχεται η Πέρασε Πέραση ψηφορία. Απορρίπτεται. 37 άρχεται η Πέρασε Πέραση ψηφορία. Απορρίπτεται. 38 άρχεται η Πέρασε Πέραση ψηφορία. Απορρίπτεται. 39 άρχεται η ψηφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 40. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 41. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 12. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 15, τροπολογία, αιτιολογική σκήψη 15, τροπολογία 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 17, 49 και 50 ταυτόσημες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Ε, Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 18, τροπολογία 51. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 21, τροπολογία 52. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Αιτιολογή σκέψη 22, τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 55, αιτιολογική σκέψη 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Ε, συγγνώμη, ε, ιδεολογική σκέψη 27, τροπολογία 6, άρχεται ψηφοφορία, πέραση πέραση Εγκρίνεται. «61, 63 και 64 μπλοκ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 66. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 67. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 68. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 69. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 70. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 71. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 74. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίες. Απορρίπτεται 75. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίες. Εγκρίνεται 76. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίες. Απορρίπτεται 77. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 78. Άρχεται η ψηφοφορία. τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 79. Άρχεται η ψηφοφορία. τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 80. Άρχεται η ψηφοφορία. τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εκρίνεται. 82, 83, 84, 85 και 86 αμπλοκ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, συγγνώμη, να τα ξαναπούμε. 82, 83 και 84 μπλοκ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 85. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 86. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 87. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου ως τροποποιήθηκε ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 41 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια στην κυρία αυτή. So, Μπορούμε να συνεχίσουμε αμέσως με την επόμενη ψηφοφορία και η επόμενη... Είναι ωραίες αυτές οι ψηφορίε, γιατί έχουμε να ζητήσουμε συμφωνίες με διάφορα νησάκια του Ειρηνικού. Και ο πρόεδρος ονειρευόταν να βρεθεί εκεί. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το σημείο 9 της σημερινής διάταξης. Συμφωνίες μεταξύ τη ευρωπαϊκή Ένωσης, ξεκινώντας ε, με την Δημοκρατία του Κυριμπάτη για την υποχρέωση θεώρηση για βραχή διαμονή. Ε, έχουμε άλλες στην Μικρονησία, του Βάλου, νήσου Σολομώντα και νήσι Μάρσαλ. Ε, κύριε Γκαμπριέλ, θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και πέρα από τα χαπόγελα θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι αυτέ οι μικρέ νησιωτικέ χώρες είναι χώρες ΑΚΕ. Άρα είτε είναι μικρέ είτε ήταν πιο μεγάλε, ε, θα πρέπει κατά την άποψή μου να του στείλουμε ένα θετικό μήνυμα σε αυτέ τι χώρε με τι οποίε γενικά θέλουμε να έχουμε μια συνεργασία. Ο Πρόεδρο, ναι, πράγματι ισχύει αυτό και επίση ε, είναι θεσμικό ζήτημα, είναι το ζήτημα των θεωρήσεων. Ε, δεν μπορούμε να γίνει, δεν μπορεί να γίνει μία ψηφοφορία για όλες τις συμφωνίες. Θα ήταν προσβλητικό προς τις χώρες αυτές να τις βάλουμε όλες μαζί, κύριε Πάτ, Μικρονησία, όλες μαζί για να ψηφίσουμε θα γίνει μια ξεχωριστή ψηφοφορία για κάθε μια από τις συμφωνίες. Γοργά όμως. Πρώτη συμφωνία που τέθηκε στη ψηφοφορία, η συμφωνία με το κύρι Μπάτι, έναρξη ψηφοφορίας. Γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι που βρίσκεται το κύρι Μπάτι. Δεν αμφέβαλα, αλλά πέρασε ψηφοφορία. Ε, συνάδελφοι, ένα της ψηφοφορίας για τη συμφωνία με την Μικρονησία. Πέρα της ψηφοφορίας. Και πάλι απαλλαγή από υποχρέωση θεώρηση για την βραχία διαμονή, ε, συμφωνία με το του βάλου. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 43 ψήφους υπέρ και 4 κατά, αποχές. Τελευταία συμφωνία για τα απαλλαγή θεώρηση που η διαπονεί για τη συμφωνία με, τους, ε, με τις νήσους Σολομόντος. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 44 υπέρ ψηφί και 4 κατάχωρες αποχές. Τελευταία συμφωνία με τις ε, νήσους Μάρσαλ. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται 43 ψήφοι υπέρ 4 κατά συγχαρητήρια στην εισηγητρία. Και έτσι, συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε την διαδικασία των ψηφοφοριών. Σα ευχαριστώ για την παρουσία σα και την υπομονή σα. Επίσης έχουμε ολοκληρώσει την ε, πρωινή πρωινό μέρο της ε, συνεδρίασή μας. Θα τα ξαναπούμε το απόγευμα ε, στις 3 η ώρα του μεσημέρι. Γεια σα.